Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Και να ξεκινήσουμε με τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Μία ανακοινώση έχω μόνο. Κυρίσω την έναρξη Τη ακρόασης των τριών επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα. Η διαδικασία γίνεται δυνάμει το άρθρο 14 του κανονισμού 2017 κάθετος 1939, βάσει το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται να διορίσουν κοινή συνενέση τον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα για μία επταετή μη ανανεώσιμη θητεία βάσει ενός καταλόγου που συγκροτεί μια Επιτροπή Επιλογής, όπως προβλέπει το ίδιο άρθρο, μετά από μια δημόσια προκήρυξη για υποβολή υποψηφιότητων. Σήμερα θα ακούσουμε ξεχωριστά σε ακροάσει του τρει επικρατέστερου υποψήφιου και θα ήθελα συνάδελφοι. Συνάδελφοι, παρακαλώ, συμπαίνουν στην αίθουσα να το κάνουν αθόρυβα. Να σα υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών έχει υποβάλει ένα σύντομο προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο τριών ερωτήσεων ε, στους υποψηφίους που απάντησαν γραπτός και έχουμε μοιράσει μάλιστα σε όλες τις γλώσσες τις απαντήσεις τους. Πριν να ρίξουμε κλήρο για τον πρώτο υποψήφιο, θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Γκρέσλε, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού που παρίστανται. Η Επιτροπή Κοντ συμμετέχει στην ακρόαση αυτή και στο τμήμα των ερωταπαντήσεων. Μάλιστα, η οργάνωση ακρόαση ακολουθεί τι αρχέ που έθεσε ο πρόεδρο Ταγιάννη στην επιστολή του τη 21η Φεβρουαρίου που σα έχουμε μοιράσει. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στην κυρία Γκρέσλε, την πρόεδρο της Επιτροπής ε, Ελέγχου του Προπολογισμού, για δύο-τρία λεπτά. Και εγώ να ευχαριστήσω. Χαιρόμαστε που έχουμε αυτή την κοινή ακρόση. Θυμίζω ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα είναι τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Για μας που είμαστε Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού είναι και Πάσχα και Χριστούγεννα. Είμαστε σε αυτό το σημείο επιτέλους που μπορούμε να επιλέξουμε το άτομο που θα παίξει αυτό το ρόλο. Άρα, μόνο ένα μπορούμε να κάνουμε, να πούμε ότι όποιος και αν επιλεγεί, το ευχόμεθα πολλή επιτυχία. Χρειαζόμαστε αυτό το θεσμό και ελπίζουμε να μπορέσει να ε, συνεχίσει την εργασία του αυτός ο τόσο χρήσιμος θεσμός με τη δική μας συμβολή. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκρέσλε. Οπότε προχωρούμε με τη διαδικασία. Θα κληρώσουμε τον πρώτο υποψήφιο για να δούμε τη σειρά των, των ακροάσεων. Εδώ στο φάκελο έχω τα ονόματα και των τριών υποψηφίων. Συναρπαστικά όλα αυτά. Θα βάλω λοιπόν το χέρι μου μέσα στο φάκελο και θα τραβήξω το όνομα του πρώτου υποψηφίου ή της πρώτης υποψήφιας. There Έχουμε τα, ονόματα τριών υποψηφίων. Διαδικαστικό εκτός μικροφώνου από την κυρία Μακοβέη. Η πρώτη ακρόαση θα γίνει με τον κύριο Αντρές Ρίτερ. Αυτός θα είναι ο πρώτος υποψήφιος. Οι υποψήφοι θα κάθονται στην άκρη του πάνελ μας. Συνήθως έχουμε τον ομιλητή μπροστά, μερικές φορές μάλλον. Ε, θα χρονομετρούμε αυστηρά και τους τρεις υποψήφιους. Θα έχουν ακριβώς τον ίδιο χρόνο για την ομιλία τους. Τους έχουμε προειδοποιήσει ότι θα είμαστε πολύ αυστηροί με το χρόνο ομιλίες και θα έχουν ακριβώς τον ίδιο χρόνο και οι τρεις. Θα ήθελα παρακαλώ να καλάσουμε τον κύριο Αντρέ Ρίτερ που θα έρθει από το πρωτόκολλο. Χρειάζεται λίγα λεπτά για να έρθει. Okay, so colleagues, um, μετά την πρώτη αυτή κλήρωση θα προχωρήσουμε με αλφαβητική σειρά. Πρώτος είναι ο κύριος Ρίτερ, μετά Μπόνερς και μετά Κοβέση. Αυτή θα είναι η σειρά. Οπότε ε, περιμένουμε δύο λεπτά για να ανέβει στο Προεδρείο ο πρώτος υποψήφιος. Έχουμε τίποτα άλλο. Εν τω μεταξύ, όσο περιμένουμε τον πρώτο υποψήφιο, να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για τη διοργάνωση της ακρόασης. Θα κάνει μια προφορική εισαγωγική ομιλία το πολύ 7 λεπτά ο κάθε υποψήφιο και μετά την εισαγωγή θα έχουμε ένα τμήμα ερωταπαντήσεων που θα κρατήσει 63 λεπτά. 14 ερωτήσεις θα θέσουν με μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, 2 τρίτα του χρόνου και 7 τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, τα 1 τρίτα του χρόνου. Ε, ένα λεπτό θα κρατούν οι ερωτήσεις και 2 λεπτά οι απαντήσεις. 3 λεπτά θα είναι τα τμήματα ερώτα απαντήσεων. Και παρακαλώ, θα είμαστε πολύ αυστηροί και εγώ και η κυρία Γκρέσλε με την τήρηση του χρόνου και θα κόβουμε το μικρόφωνο των ομιλητών. Αλλιώς δεν θα προλάβουν να θέσουν όλες τις ερωτήσεις τους. Κύριε Σόγκορτ, έχετε διαδικαστικό ή απλώς θέλετε το λόγο. Έχουμε κατάλογο, καταρτίζουμε κατάλογο ομιλητών. Έχουμε και διερμηνία, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη μητρική σας γλώσσα επειδή όμως υπάρχει διερμηνία, δεν χρειάζεται να μιλάτε με αστρονομική ταχύτητα για να σας προλαβαίνουν και διερμηνείς. Περιμένουμε τον πρώτο μας υποψήφιο. Πού είναι? Έρχονται από την αίθουσα αναμονή ε, στο πρωτόκολλο. Χρειάζεται λίγα λεπτά λοιπόν για να έρθουν μέχρι το κτίριο αυτό. Παρακαλώ, λίγη υπομονή. Θα έρθουν ανα πάσα στιγμή υποψήφια. Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, περιμένοντα ε, τον υποψηφιό μας, ε, τον πρώτο υποψηφιό μας, τον κύριο Αντρέ Ρίτε, να καθίσει και να νιώσει άνετα. Ε, παρακαλώ λίγο σεβασμό προς τους υποψηφίους. Ήρθε ο υποψηφιός μας και περιμένει να κάνει την ομιλία του. Οπότε δεν είναι σωστό να μένουν όρθιοι κάποιοι στην αίθουσα. Παρακαλώ, καθίστε. Ο κύριος Αντρέ Ρίτερ είναι ο πρώτος μας υποψήφιος. Θα έχει 7 λεπτά για να μας κάνει την εισαγωγική του ομιλία. Παρακαλώ, προσοχή στο χρονόμετρο, κύριε Ρίτερ, γιατί όταν ε, λήξει ο χρόνος πρέπει να σταματήσετε. Θα σα θέτουν ερωτήσει που θα κρατούν ένα λεπτό και εσεί θα έχετε δύο λεπτά για να απαντάτε. Όλα αυτά θα τηρήσουμε πολύ αυστηρά για όλου του υποψηφίου. Γι' αυτό το μάτι σα στο χρονόμετρο. Αν είστε έτοιμο και αν είμαστε όλοι έτοιμοι, θα ξεκινήσουμε με την πρώτη επτάλεπτη ομιλία του κυρίου Ρίτερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Παρόλο που φαίνεται προφανές, το κύριο ερώτημα είναι γιατί χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή με άλλα λόγια ε, από πού ερχόμαστε χωρίς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προς τα πού δεύουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η απάτη και η διαφθορά εις βάρος ε, του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θίγει τους οικονομικούς πόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκαλεί ζημία. Βέβαια γνωρίζετε ότι έχει και μια ευρύτερη διάσταση. Η απάτη και η διαφθορά αποδυναμώνουν την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μάτια των φορολογουμένων. Εξού και η ανάγκη για μια ισχυρή προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Κάτι τέτοιο είναι ζωτική σημασία. Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που εξηγούν γιατί η ποινική δίωξη στην προστασία οικονομικών συμφερόντων δεν ήταν τόσο αποτελεσματική όσο θα γινόταν. Συνδέονται και οι τρεις λόγοι με το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η δίωξη ακολουθούσε μια εθνική προσέγγιση. Καταρχήν, η πολιτική για τις ποινικέ διώξεις και την ποινική έρευνα ήταν κατακαιρματισμένη και παρά τα επιτεύγματα Μία εθνική προσέγγιση δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Ω εκ τούτου θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα να έχουμε μια ευρωπαϊκή εισαγγελία που θα δικαιούται να διαμορφώνει και να εφαρμόζει τη δική τη πολιτική για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων και την ποινική δίωξη. Και σημαίνει μια νέα πανευρωπαϊκή προσέγγιση από μια πανευρωπαϊκή σκοπιά. Και κάτι τέτοιο θα υλοποιηθεί μόνο αν έχουμε μια πλήρω ανεξάρτητη ευρωπαϊκή εισαγγελία. Δεύτερον, τα εθνικά δικαστικά συστήματα δεν ήταν και πολύ πρόθυμα με την ε, ε, διερεύνηση και δίωξη διασυνοριακών εγκλημάτων. Περιοριζόταν μόνο στις εθνικές πτυχές τέτοιων αδικημάτων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μία ενιαία υπερεθνική εισαγγελία είναι απαραίτητη, γιατί θα είναι ικανή να έχει μια γενικότερη επισκόπηση της κατάστασης και άρα να διενεργεί πιο συνολικές ε, έρευνες. Ε, τρίτον, ένας πρακτικός λόγος ε, για τις ανεπαρκείς έρευνες σε θέματα οικονομικών συμφερόντων ήταν η έλλειψη πόρων σε εθνικό επίπεδο. Η εμπειρία από τα οικονομικά εγκλήματα μας διδάσκει ότι οι πόροι είναι ανεπαρκείς για να αντιμετωπίσουν περίπλοκες ε, αξιόπινες πράξεις και εγκληματική δραστηριότητα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας αποτελεσματικά, να συγκεντρώσουμε τις ικανότητές μας να δημιουργήσουμε συνέργειες και να θεσπίσουμε καλή συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους. Και σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βασικοί ενδιαφερόμενοι είναι η Olaf, η Eurojust και η Europol. Συνέργειες με αυτά τα σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αυτούς τους φορείς ε, θα προέρχονται από συμφωνίες για, για συνεργασία. Και φυσικά θα πρέπει να τα προσδιορίσουμε όλα αυτά και σχέση με την ΟΛΑΦ είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί η ΟΛΑΦ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν συμπληρωματικού ρόλου. Είναι οι δύο του ίδιου νομίσματο. Αυτό βέβαια δεν υποτιμά το σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσουν η Eurojust και η Europol στα πλαίσια των εντολών του για να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εν όψη λοιπόν της αποτελεσματικής χρήση των πόρων που σας ανέφερα, ε, είναι κέρια σημασίας η σχέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με όλα τα με όλους αυτούς τους φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχει ούτε επικαλύψεις, αλλά να μην αφήνει και κενά ταυτόχρονα. Και παρά τον υπερεθνικό της χαρακτήρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στηρίζεται στη συνεργασία με τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη, κυρίως σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που θα παρέχουν οι εθνικές αρχές η ομαλή, γρήγορη και αξιόπιστη ροή και ανταλλαγή πληροφοριών θα έχει κρίσιμη σημασία για το έργο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Σε ό,τι αφορά τις μη συμμετέχουσες χώρες μέλη, ε, έχω αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλή συνεργασία περιπτωσιολογικά και το καθεστώς που προβλέπει ο κανονισμός διευκολύνει τέτοιου είδους συνεργασία. Κατά τη γνώμη μου βέβαια, ένα ειδικό πλέγμα νομικών εργαλείων με αυτά τα κρατημέλη θα εξασφαλίσουν ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια δικαίου. Σε ό,τι αφορά την εσωτερική οργάνωση της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η διαδικασία λήψη αποφάσεων είναι αρκετά περίπλοκη. Και αυτό είναι αναμφισβήτητο. Γι' αυτό ο Ευρωπαϊκός Γενικός Εισαγγελέας, έχει το καθήκον μαζί με το Συλλογικό Όργανο των Εισαγγελέων να εξασφαλίσει μια ομαλή και ταχύτητα διαδικασία. Θα πρέπει να είναι σαφείς καθορισμένες ε, και εύχριστες οι οι διαδικασίε και ο εσωτερικό κανονισμό. Γιατί σίγουρα ο Ευρωπαίο Γενικό Αγγελέα θα είναι η κινητήριο δύναμη για μια ε, εύρυθμη μεθοδολογία και πρακτική. Σε ό,τι αφορά τις διάφορες περιπτώσεις αμοιβέ και έγκαιρες ανταλλαγές πληροφοριών είναι σημαντικοί με τα τμήματα, τα μόνιμα και τους εντεταλμένους ε, εισαγγελείς. Και αυτό ισχύει πολύ περισσότερο ε, που υπάρχει το ενδεχόμενο πολλοί Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς να επιλαμβάνονται ταυτόχρονα τις ίδιες διασυνοριακές υποθέσεις. Επίσης, ε, η συγκρότηση, σύσταση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας συνιστά ένα τεράστιο βήμα πρόοδου. Επιπλέον, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, όχι το μοναδικό όμως, σε ένα τελείως νέο νομικό τοπίο σε ό,τι αφορά την προστασία οικονομικών συμφερόντων. Και για να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας προς τον Ευρωπαίο Φορολογούμενο, η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας θα εξαρτηθεί από το πώς θα συμπεριληφθεί και θα συνεργαστεί στα πλαίσια αυτού του νέου πλαισίου. Τέλος, η λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν περιορίζει την, την ανεξαρτησία του, αλλά είναι εχέγγυο της ανεξαρτησίας αυτής. Επίσης, να σας παρουσιάσω την άποψη ενός αγγελέα για την έννοια που έχει μια καλή και αποτελεσματική δίωξη. Πιστεύω ότι οι εισαγγελείς θα πρέπει να είναι οι θεματοφύλακες του νόμου η αξιοπιστία τους και η συνέπειά τους ε, ε, απορρέει από την προσήλωσή τους στο κράτος δικαίου. Ως εκ τούτου, καλή και αποτελεσματική δίωξη σημαίνει ε, πιστό σεβασμός και αυστηρό σεβασμός των δικονομικών εγγυήσεων και των μεμονωμένων δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται και στο ρωσιακό δίκαιο και στις εθνικές ένωμες τάξεις. Σας ευχαριστώ. κοιτάξτε, ήσασταν ο πρώτος. Δεν ήθελα να σας διακόψω, αλλά Πήγε κάποια αναταρχή στην αίθουσα και σα ζητώ συγγνώμη. Ελπίζω πραγματικά οι συνάδελφοι να μην πηγαίνουν μπρο πίσω. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ακρόαση, είναι και συνέντευξη για πρόσληψη. Πρέπει να σεβαστούμε του υποψηφίου. Λοιπόν, ε, σημειώνω λοιπόν και θέλω να μπει στα πρακτικά. Δεν ήθελα να σα διακόψω γιατί θα μπορεί να ήταν χειρότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω πω ήταν εύκολη η καταστροφή για σα. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σα και τώρα να περάσουμε ευθύ στι ερωτήσει. Η κυρία Μετσόλα πλευρά του ΕΛΚ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Ρίτερ για την παρουσίασή σα. Πείτε μας λίγο περισσότερα για την πείρα σας, για την αντιμετώπιση ε, υποθέσεων ε, μεγάλης δημοσιότητας. Γιατί ο εισαγγελέα, ο Ευρωπαίος εισαγγελέα θα πρέπει να αντιμετωπίσει μερικές τέτοιες υποθέσεις που θα είναι ιδιαίτερα δυσχερείς και πολύ προβεβλημένες. Έχουμε δει διάφορες περιπτώσεις όπου διάφοροι εισαγγελείς αρνούνται να αναλάβουν δράση, αρνούνται ούτε καν να κάνουν ανακρίσεις να αρχίσουν να εξετάζουν υποθέσεις. Πώς θα συνεργαστείτε εάν κάποια κράτη-μέλη δεν είναι συνεργάσιμα. Και δώστε μας μερικά παράδειγματα μεθόδων που χρησιμοποιούν οι εγκληματικέ οργανώσεις για να, ε, ε, ε, βγάλουν, για να βγάλουν λεφτά και να κάνουν απάτε σε βάρος του προπολισμού της Ένωσης. Δύο λεπτά κύριε Ρίτερ. Ναι είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα αυτό που θέτεται. Όπως είπα, ο ρόλος ενός εισαγγελέα είναι να ε, τηρεί αυστηρά ε, τις αρχές της νομιμότητας. Όταν ε, ε, ενημερωθεί ότι υπάρχει ενδεχόμενο παράνομης πράξη πρέπει να παρέμβει τι στήριξη θα λάβει. Αυτό εξαρτάται από τη δομή του οργανισμού στον οποίο ανήκει. Το γεγονός ότι ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας έχει την απαραίτητη ανεξαρτησία και έχει τις αναγκαίες αρμοδιότητες που ε, προκύπτουν από την ευρωπαϊκή φύση του θεσμού μας επιτρέπει, πιστεύω, και στην πράξη και σε περιπτώσεις ε, που έχουν υψηλή δημοσιότητα να διώκονται ε, τα ενδεχόμενα ε, εγκληματικών πράξεων. Τώρα, αν υπάρχει αντίδραση από κάποιο κράτος μέλος ε, για να υποστεί δίωξη, πρέπει να δούμε. Αλλά πιστεύω ότι εκεί θα βοηθήσει και η στήριξη του Κοινοβουλίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι παρόν και ο εισηγητής του Κοινοβουλίου. Αλλά ναι μεν ήμασταν ανεξάρτητοι, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς στα πλαίσια της νομιμότητας μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου υπήρξε πολύ κριτική στην δημοσιότητα. Όμως ε, το βασικό είναι ότι εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε τον Ευρωπαίο φορολογούμενο και επειδή πολλές φορές ε, μπορεί οι κατηγορούμενοι να είναι και δημόσια πρόσωπα και εκπρόσωποι πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί όσον αφορά την τήρηση της αρχής νομιμότητας. Με συγχωρείτε πρέπει να σας ε, διακόπτω. Είναι η πρώτη προειδοποίηση που σας δίνω, να μην υπερβαίνετε το χρόνο σας. Δεύτερη ερώτηση. Η κυρία Ζίπελ, σοσιαλιστές. Κύριε Ρίτερ, με τι τρόπο θα σεβαστείτε όλες τις ε, απαιτήσεις που χρειάζονται όπως αναφέρει το άρθρο 14 του κανονισμού και συγκεκριμένα είναι σίγουρη ανεξαρτησία σας πέραν ε, αμφιβολίας. Έχετε τα αναγκαία προσόντα για να αναλάβετε αυτήν την υψηλότερη εισαγγελική αρχή όπως θα μπορούσατε να κάνετε και κράτη-μέλη. Και από πότε ε, έχετε τα αναγκαία προσόντα. Δύο λεπτά κύριε Ρίτερ. Ε, κοιτάξτε, εκτός του γερμανικού σύστηματος δεν μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς ε, την απάντησή μου. Η προπόθεση ανεξαρτησίας υπάρχει από τη στιγμή που αναλαμβάνουμε υπηρεσία. ο εισαγγελέα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ε, είναι υπόλογο μόνο έναντι του νόμου. Αυτό είναι προπόθεση ευθύ εξ αρχή. Δεν υπάρχει κανένα ε, ιδιαίτερο έλεγχο, εάν και κατά πόσο ασκεί ανεξάρτητα κανεί τα καθήκοντά του. Είναι βέβαια αναγκαίο από την πράξη. Αυτό, που μπορώ να πω για, αυτό μπορώ να πω την ανεξαρτησία. Για τι άλλε προποθέσει που, που καθορίζονται για αυτό το υψηλό αξίωμα, πρέπει κανεί να έχει τα αναγκαία προσόντα Στη Γερμανία υπάρχουν διάφορες εξετάσεις και περίοδοι ε, ελέγχου από ανώτερες αρχές που πιστοποιούν ότι έχει τις αναγκαίες ικανότητες ε, διοίκησης ε, για να μπορεί να ηγείται μια υπηρεσία. Αυτά είναι θέματα που κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου απέδειξα ότι τα διαθέτω. Για την ανεξαρτησία θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντική για μένα και είμαι και μέλος της ε, Διεθνούς Ένωσης ε, Δικαστών που εργάστηκε για ε, διεθνή θέματα και συγκεκριμένα για, εργάστηκα σε μια επιτροπή αυτού του Διεθνούς Οργανισμού που ασχολείται με την ποινική δικονομία και το ποινικό δίκαιο. Και μου τέθηκαν ερωτήσεις για την κατάσταση στην Πολωνία και εκφράστηκα από αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. η κυρία Χέλγα Στίβεν. Ένα λεπτό. My apologies, she's not here. Α, συγγνώμη, δεν είναι εδώ η κυρία Χέλγα Στίβεν. Η κυρία Χάουσμανούβα από την Άλντε. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Μία ερώτηση. Με βάση τις γραπτές απαντήσεις που δώσατε οι μελλοντικέ σα σχέσει μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Αγγελία και των κρατών μελών που δεν θα συμμετέχουν. Πώ ε, θα αξιοποιήσετε τι δυνατότητε που έχετε να ε, βοηθηθείτε από τους εθνικούς ανταποκριτές του Eurojust. Eurojust. Είναι κάτι, ο θεσμός αυτός που δημιουργήθηκε πρόσφατα για να ενθαρρύνουν ε, τα κράτη αυτά που δεν συμμετέχουν να ενταχθούν στο θεσμό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και για να υπάρχει συνεργασία. Και δεύτερον, η εργασία τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μία από τι ανησυχίε μα κατά την ε, συζήτηση του κανονισμού για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα ήταν ότι δεν θα ήταν απόλυτα ευρωπαϊκή η αρχή αυτή. Ότι τα εθνικά συμφέροντα θα καθόριζαν τη στάση των εντεταλμένων εισαγγελέων. Τι συγκεκριμένα μέτρα λοιπόν θα πάρετε για να εγγυηθείτε τη δημιουργία ενό ανεξάρτητου σώματο, μια ε, ανεξάρτητη και πραγματικά ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ευχαριστώ. Ρίτα, παρακαλώ, δύο λεπτά. Για την πρώτη ερώτησή σας. Σχέση με τα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν στο θεσμό μου και σχέση με το Eurojust. Ο ρόλος του Eurojust είναι πολύ σημαντικός. Αυτό ισχύει. Βεβαίω η Eurojust δεν έχει τι αρμοδιότητε με τον εισαγγελέα. Αλλά εάν υπάρξει ένα τέτοιο οικονομικό έγκλημα στα κράτη-μέλη που δεν ε, συμμετέχουν, με βάση τον κανονισμό και του Eurojust και τον κανονισμό της ε, εισαγγελία μπορούν να συνεργαστούν. Το Eurojust θα πρέπει να εμπλέξει και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να υπάρχει μια κοινή ομάδα ερευνών. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σε αυτέ τι περιπτώσει, σε αυτέ τι υποθέσει για να ε, προστατευτούν πλήρω τα οικονομικά συμφέροντα τη Ένωση. Αλλιώ θα υπήρξε προφανώ, θα υπάρξει προφανώ μια, ένας κατακαιρματισμός. Πρέπει λοιπόν να συμμετάσχει και το Eurojust. Πρέπει να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πιστεύω ότι έτσι μπορεί να συμβάλλει πολύ, ούτως ώστε να υπάρχει ουσιαστική συνεργασία και με τα μη συμμετέχοντα κράτη-μέλη. Και τώρα, η ανεξαρτησία των κρατών μελών, στα κράτη-μέλη τα ίδια. Αυτό είναι ένα μεγάλο καθήκον. Θα πρέπει να κάνει διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη Ευρωπαίου Εισαγγελές για να επιτύχουμε αυτή την ανεξαρτησία. Η δυνατότητα που έχουμε να αντικαταστήσουμε τον ε, εντεταλμένο με κάποιον άλλον Αλλά βεβαίως και αυτοί οι συνάδελφοι θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και να τηρούν αυστηρός τα αναγκαία κριτήρια που καθορίζει ο κανονισμός. Ευχαριστώ πολύ. Η Εύα Ζολή για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ρίτερ, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Στην δομή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας έχετε κάποια τμήματα με εθνικούς εισαγγελείς που θα είναι επιφορτισμένοι με έρευνες που αφορούν κάποιο κράτος ή θα ανατίθεται η έρευνα σε έναν εντεταλμένο Ευρωπαϊκό Ευρωπαίο εισαγγελέα. Τι θα γίνει σε περίπτωση που ο συγκεκριμένο εντεταλμένο ε, εισαγγελέα αποφασίσει να μην λάβει δράση. Και δεν είναι θεωρητική μόνο η περίπτωση, γιατί και στην πατρίδα μου δυστυχώ έχουμε την παράδοση οι εισαγγελείς να πρόσκειται στην εξουσία και να μην αναλαμβάνουν πρόθυμα δράση. Κύριο Ρίτερ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Γιατί και εγώ θέτω στον εαυτό μου αυτό το ερώτημα από τότε που ασχολούμαι με το θέμα του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα. Τι δυνατότητε υπάρχουν εάν ένα εντεταλμένο εισαγγελέα για οποιοδήποτε λόγο δεν δρά με βάση την εντολή που του έχει ε, δοθεί. Πρέπει να επιλεγούν ε, εισαγγελείς οι οποίοι να θέλουν να συνεργαστούν. Αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, προβλέπεται δυνατότητα στον κανονισμό ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας της ε, αντίστοιχης χώρας να αναλάβει την έρευνα. Αυτό σημαίνει επιπλέον φόρτο εργασίας για το σύστημα. Αν προκύψει κάτι το καλύτερο, το βέλτιστο θα ήταν η πίεση που θα ασκηθεί να οδηγήσει στο καλό αποτέλεσμα. Η πίεση που μπορεί να ασκήσει ένας γενικός εισαγγελέα στα κράτη-μέλη να οδηγήσει στην ανάληψη δράσης από τα κράτη-μέλη. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω ούτε εγώ Πώ συγκεκριμένα θα εξελιχθεί μια τέτοια κατάσταση, τι ρύθμιση μπορεί να βρεθεί. Να βρεθεί. Πρέπει να ε, επιχειρήσουμε να συμφωνήσουμε με το κράτος μέλος, ε, ενδεχομένως να αντικατασταθεί αυτός ο εισαγγελέας, αν αυτή είναι η καλύτερη λύση. Και αν δεν είναι δυνατόν, τότε ο Ευρωπαίος εισαγγελέας της αντίστοιχης χώρας να αναλάβει αυτή την έρευνα με ε, τις δυσχέρειες που θα προκύψουν βέβαια γιατί θα πρέπει να κάνει την έρευνα εξ αποστάσεως. Ευχαριστώ κύριο Ράντεφ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, έχετε μια πραγματικά εντυπωσιακή σταδιοδρομία πίσω σας. Φαίνεται από το βιογραφικό σας ότι έχετε αποκομίσει μεγάλη εμπειρία εθνική σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Σίγουρα θα έχετε χειριστεί και ευαίσθητε υποθέσει που συμπεριλάμβαναν και την απάτη με ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτά θα είναι και το, η δουλειά σα σε καθημερινή βάση ω Ευρωπαίου εισαγγελέα. Και θα πρέπει βεβαίω να εξασφαλίζετε ότι θα σημειώνετε πρόοδο. Μπορείτε να μα δώσετε λοιπόν ένα παράδειγμα υπόθεση που έχετε χειριστεί και που συμπεριλάμβανε την κατάχραση Ευρωπαϊκή παϊκών κονδυλίων και πώς ακριβώς ανταποκριθήκατε στις προσδοκίες της κοινή γνώμης και του τύπου. Επίσης, τι πιστεύετε για τη μελλοντική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κύριε Ρίτε. Να ξεκινήσω με το δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σας. Όπως είπα και εισηγητικά, είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι η ισχυρή προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο αν υπάρχει μια πανενωσιακή, πανευρωπαϊκή προσέγγιση. Αν υπάρχει δηλαδή μια αρχή εισαγγελική η οποία θα έχει στη διάθεσή της του απαραίτητους πόρους και η οποία θα μπορεί να διατυπώνει μια κοινή ε, και ομοιόμορφη στρατηγική για το πώς θα αντιμετωπίζεται ένα φαινόμενο το οποίο θα είναι πανευρωπαϊκό. Αν με ρωτάτε ποια ήταν η μεγαλύτερη υπόθεση στην οποία εγώ συμμετείχα. Δεν μπορώ φυσικά να σας τα αποκαλύψω όλα, ε, γιατί είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει τελεσιδικήσει ακόμη. Μπορώ όμως να σας πω ότι πρόκειται για μια υπόθεση στην οποία λόγω μιας τεχνητής, ε, ενός τεχνητού διαχωρισμού ενός έργου ε, παρακάμφθηκαν ευρωπαϊκές απαιτήσει. Υπόθεση στην οποία ε, προκλήθηκε μια ζημία ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ. στην οποία ενδέχεται μάλιστα να εμπλέκονται και πολιτικοί, άνδρες και γυναίκες. Διεξήγαμε λοιπόν τις, έρευνες, τις έρευνές μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, με συμμετοχή μάλιστα και του Όλαφ. Καταλήξαμε λοιπόν στην απόδοση κατο... κατηγοριών. Ε... Έγινε μια, ε, η εκδίκαση σε πρώτο βαθμό της υπόθεσης. Βρισκόμαστε στο στάδιο της έφεσης αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Η κυρία Κινίτση για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Η σχέση ανάμεσα στην εκτελεστική εξουσία και την εισαγγελική αρχή ε, ρυθμίζεται με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κράτη-μέλη. Με ποιον τρόπο λοιπόν εσείς θα προωθήσετε τον προδραστικό ρόλο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα στον εντοπισμό και τη διερεύνηση ε, αδικημάτων κατά της, ε, των οικονομικών συμφερόντων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης με ομοιόμορφο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Και πώς ακριβώς θα εξασφαλίσετε ότι η απέτηση ανεξαρτησίας υπό το άρθρο 6 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συγγελία θα εξασφαλίζεται σε όλα τα επίπεδα ε, λειτουργίας και δράσης ε, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. θεωρώ ότι δικαίως αναφέρεστε σε αυτή την απέτηση ανεξαρτησία, Είναι το βασικό, το ουσιώδες στοιχείο ε, ώστε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το έργο της να στεφτούν με επιτυχία. Γιατί χωρίς ανεξαρτησία δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους της. Είπα άλλωστε και εισαγωγικά, γιατί πιστεύω ότι η ανεξαρτησία αυτή εξασφαλίζει ε, την ομοιόμορφη, ενιαία ε, στάση και πολιτική που θα τηρήσει αυτή η εισαγγελική αρχή. Αν κατάλαβα σωστά το ερώτημά σας, θέλω να σας απαντήσω λέγοντας ότι το ερώτημα είναι πώς ο εντετελμένος Ευρωπαίος εισαγγελέα θα ανταποκρίνεται στα ίδια ε, κριτήρια ανεξαρτησίας. Νομίζω ότι ο κανονισμός απαντά ε, καθώς παραθέτει και περιγράφει τις προϋποθέσεις που θα πρέπει κάποιος να εκπληρώνει ώστε να μπορεί να επιλεγεί ως ευρω... εντεταλμένος Ευρωπαίος εισαγγελέα. Για μην ξεχνάμε ότι ο Ευρωπαίος Γενικός εισαγγελέα θα είναι εκείνος ο οποίος σε συνεργασία με το σώμα των εισαγγελέων θα διαλέγουν εκείνους που θα κομίζουν τα περισσότερα εχέγγυα ανεξαρτησίας. Άρα ενεργά θα συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην επιλογή του καλύτερου δυνατού προσώπου προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία της διαδικασίας. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο ισχυρότερος δυνατός μηχανισμός τον οποίο μπορεί να θεσπίσει κανείς προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία των ε, εισαγγελέων, των υποψηφίων σε μια πρώτη φάση που θα κληθούν να ε, χειρίζονται τις ε, εκάστοτε υποθέσεις. Ευχαριστώ. Έφτασε και η κυρία Στίβενς, οπότε θα της δώσω το λόγο για να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ε, τώρα ε, να δώσω το λόγο στην κυρία Μακοβέη από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές. Ε, Ευχαριστώ. Μια και μιλάτε γερμανικά, θα μιλήσω και εγώ τη δική μου μητρική γλώσσα. Είδα στο βιογραφικό σας ότι τα τελευταία 8 χρόνια βρίσκεστε σε, έχετε αναλάβει ηγετικέ θέσει. Μπορείτε να μα δώσετε κάποιε πληροφορίε σχετικά με τι εμπειρίε που έχετε συγκεντρώσει στη διαχείριση, στη διοίκηση. Πόσου υφισταμένου είχατε, τι προπολογισμό ε, είχατε στη διάθεσή σα και χειριστήκατε. Δεύτερο ερώτημα. Θα μπορούσατε να μας δώσετε ενδεχομένως κάποιες, ε, κάποια παραδείγματα υποθέσεων απάτης κατά ευρωπαϊκών κονδυλίων τις οποίες χειριστήκατε εσείς, αλλά που να έχουν τελεσιδικήσει, που να έχει ληφθεί πλέον οριστική απόφαση. Επίσης, πώς ε, αντιμετωπίσατε, αν ε, έτυχε να, σας, ε, αν, να αντιμετωπίσετε και τέτοια, την πολιτική πίεση που ενδεχομένως σας ασκήθηκε. Να ξεκινήσω με το τελευταίο ερώτημα σας, κυρία Μακοβέη. Πολιτική πίεση, δόξα το Θεό, λέω, δεν έχω ζήσει ποτέ. Δεν μου έχει ασκηθεί ποτέ τέτοια πολιτική πίεση. Και είμαι ευγνώμων, πρέπει να σας πω, για το γεγονός ότι κατάφερα να επιτελέσω το έργο μου ως εισαγγελέα χωρίς τέτοια πολιτική πίεση. Κριτική μου ασκήθηκε, αλλά δεν ήταν κριτική την οποία, ε, την οποία θα μπορούσα να την εξισώσω με εκείνη που ασκείται σε εισαγγελίε σε άλλες χώρες. Και φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Εγώ λοιπόν είμαι επικεφαλής ε, μιας εισαγγελικής αρχής που αυτή τη στιγμή έχει 127 ε, υπαλλήλους. Τον προπολογισμό μας δεν μπορώ να σας τον αποκαλύψω δυστυχώς, διότι είναι αρμοδιότητα άλλης μονάδας Μπορώ όμως να σας πω ότι τα τελευταία 14 χρόνια ε, έχω θητεύσει σε επιτελικές θέσεις και αυτό που έχω μάθει από την εμπειρία μου αυτή είναι το πόσο σημαντικό είναι να εκτιμάτε και να γίνεται σεβαστό βεβαίω το έργο των υφισταμένων σου, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να λειτουργεί κανείς και ως πρότυπο παράδειγμα προς μίμηση, γιατί ε, το έργο μιας εισαγγελίας είναι συλλογικό και νομίζω ότι το έργο μας έχει στεφθεί με επιτυχία το έργο της υπηρεσίας της οποίας έχω ηγηθεί αφορούσε ε, και δύσκολα θέματα όπως η κυβερνοασφάλεια, ε, τρομοκρατία. Θα ήθελα να σας απαντήσω ε, εκτενέστερα και να σας δώσω και περισσότερες πληροφορίες, αλλά δυστυχώς τέλειωσε ο χρόνος μου. Ευχαριστώ η Ingeborg Γκρέσλε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το βιογραφικό σας. Νομίζω ότι όλοι οι υποψήφοι έχουν εντυπωσιακό βιογραφικό. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ε, τι εμπειρίες είχατε στη συνεργασία σας με τον Όλαφ στην καταπολέμηση υποθέσεων απάτης. Είπατε και εισαγωγικά και σας ευχαριστώ ότι μόλις το 50% των υποθέσεων του Όλαφ τελικά εκδικάζονται στα εθνικά δικαστήρια και σας ευχαριστώ που το ε, είπατε γιατί ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να θεσπίσουμε αυτήν την ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί αυτό. Ποια είναι λοιπόν η δική σας εντύπωση όσον αφορά τη συνεργασία σας με τον Όλαφ, αυτή την αρχή εν γέννη είναι κατάλληλη για την καταπολέμηση των περιπτώσεων ε, απάτης. Τι, τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε. Ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Είναι σημαντικό το ερώτημα που θέτετε. Και είναι ερώτημα που συνδέεται και με την αναδιατύπωση του κανονισμού του Όλαφ. Με τον Όλαφ, εμείς ως Γερμανική Εισαγγελία είχαμε πάντοτε μια πολύ καλή συνεργασία. Αποφασιστική σημασία για εμάς είναι το εξή: Ο Όλαφ έχει μακροχρόνια εμπειρία πώς μπορεί κανείς να χειρίζεται και να αξιολογεί αυτέ τι αυτές τις υποθέσεις και από την άποψη του ευρωπαϊκού, του ενωσιακού δικαίου διότι πολλές φορές η στάση μας εξαρτάται και από την διοικητική αξιολόγηση. Το αν κάτι είναι, αντίκειται λοιπόν στο κοινοτικό δίκαιο, εκεί μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ ο Όλαφ. Θέλω να πω ότι ακόμη και αν ε, οι στόχοι συγκλίνουν και, οι εργασίες, και ταυτόχρονα οι εργασίες εκτελούνται σε διαφορετικά επίπεδα, υπάρχει ένας καλός συντονισμός, μια καλή συνεργασία και η εμπειρία του Όλαφ είναι πάντοτε ύψης της σημασίας για μας. Αν λοιπόν αυτές τις δυνατότητες του Όλαφ μπορέσουμε να τις αξιοποιήσουμε με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμοστούν πλήρως και στις ποινικέ διαδικασίες, πραγματικά θα έχουμε κερδίσει πάρα πολλά. Ξέρω ότι διεξάγεται και μια τέτοια συζήτηση για το πώ μπορούν να αξιοποιούνται και στοιχεία στα οποία, ή ενδείξει, αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία συλλέγει ο Όλαφ στι εθνικέ δικαστικέ διαδικασίε που ακολουθούνται. Τώρα το πώ τι τελική μορφή θα πάρουν όλα αυτά, δεν μπορώ να σα το πω εγώ. Όμω είναι πραγματικά εξαιρετική προπόθεση το να έχουμε αυτήν την υποστηρικτική διαδικασία του Όλαφ. Και για να γίνει αυτό χρειάζονται φυσικά διαδικαστικά και δικαστικά εχέγγυα. Αν υπάρχουν τέτοια εχέγγυα προκειμένου να μπορούν τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγει ο να αξιοποιούνται σε εθνικό επίπεδο από τα δικαστήρια, τότε βεβαίω αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ θα το υποστηρίξω. Σα ευχαριστώ. Κυρία Τάνια Φαγιόν, για τους σοσιαλιστές. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Ασχοληθήκατε ποτέ με περίπλοκα διασύνοριακά θέματα, με περίπλοκες ε, διασύνοριακές ε, έρευνες. Δυστυχώς δεν λειτουργεί πια το μικρόφωνο της κυρίας Φαγιού. The microphone. Oh, uh, yes? Okay, <laughs> sorry.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 and Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πώς θα αποδείξετε την... Ε, πώς θα ε, πείσετε τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ε, συμπεριληφθεί ακόμη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να το κάνουν σε ένα μεταγενέστερο επίπεδο και ασχοληθήκατε ποτέ με περίπλοκες διασυνοριακές ε, έρευνες που εμπερίχαν και σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ εθνικών δικαστηρίων. Κοιτάξτε, το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας ε, έχει πολιτική φύση. Δεν θα πω πολλά. Αλλά το πόσο μπορεί να ασκήσει πειθό το λειτουργήμα του εισαγγελέα είναι σαφές, συμφωνώ. Βεβαίως. Καλύτερα να πείθει κανείς, να είναι τμήμα των ε, μέσων που διαθέτει για να κάνει τη δουλειά του. Έχω συμμετάσχει σε έρευνες ε, πολύ σοβαρών διασυνοριακών αδικημάτων που αφορούσαν την Ιταλία, την Τσεχία και τη Γερμανία. Υπήρχαν ε, υποθέσεις αφάτης, απάτης ΦΠΑ διασυνοριακού χαρακτήρα. Μαζί με την Eurojust ε, ε, συστήσαμε μια κοινή ομάδα ερευνών και συγκρίνω την ε, εργασία μιας τέτοιας ομάδας υπό την, υπό την αιγίδα του Eurojust και τι θα μπορούσε να κάνει μια κοινή μελέτη υπόθεσης υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και θεωρώ ότι μπορεί να κάνει περισσότερα. Ο συντονισμός θα είναι με πολύ λιγότερες ε, τριβές. Ο συντονισμός θα είναι πολύ πιο απλός από τη φάση των ερευνών αν μπορούν να συνεργαστούν δύο εισαγγελίες από κοινού. Όχι μέσω ε, της νομικής βοήθειας. Βεβαίως είναι καλύτερο να υπάρχει ένας ε, συντονισμός τουλάχιστον μέσω της Eurojust. Είναι πολύ εύκολο να ανταλλαγούν στοιχεία έτσι και πολύ πιο γρήγορα. Ήδη και η Eurojust ε, βοήθησε σε αυτή την ε, περίπτωση και υπήρξε καταδίκη με πολύ ψηλό πρόστιμο. Αλλά το αποτέλεσμα που επετέφθη σε μία χώρα μετά πρέπει να μεταφερθεί στις άλλες. Ε, υπάρχουν γλωσσικά προβλήματα, πρέπει να γίνουν μεταφράσει. πρέπει να ασχοληθεί η άλλη χώρα με βάση το δικό τη σύστημα. Αν έχουμε δύο συναδέλφου που συνεργάζονται και που τα αποτελέσματα μπορούν να μπουν σε μία διαδικασία, αυτό ε, είναι μεγάλο κέρδο από πλευρά χρόνου και αποτελεσματικότητα σε σχέση με την κλασική μορφή συνεργασία τη νομική βοήθεια. Ακόμη και γίνεται στα πλαίσια μια ε, κοινή ομάδα έρευνα. Ευχαριστώ πολύ. Και τέλος, η Χέλγα Στίβενς από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, που είναι μέλος της ομάδας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών ECR. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, γιατί με πρόλαβε η κυρία Εύα έθεσε την ίδια ερώτηση που είχα προετοιμάσει κι εγώ. Εντάξει. Οπότε περνάμε σε ερωτήσει των μελών τη Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Ευχαριστώ. Να επανέλθω στο θέμα τη Όλαφ. Στην αρχή είπατε ε, γιατί οι εθνικές αρχές σε αυτά του τουλάχιστον που βλέπετε δεν δίνουν πολύ συνέχεια στις έρευνες της Όλαφ. Οπότε το ερώτημά μου είναι τι ρόλο βλέπετε να έχει η Όλαφ για διοικητικές ε, για παράδειγμα υποθέσεις, όταν θα αρχίσει να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διότι οι διαδικασίες είναι διαφορετικές. διότι οι διοικητικές έρευνες μπορεί να είναι ιδιαίτερα περίπλοκες. Πώς μπορείτε να συνεργαστείτε λοιπόν σε τέτοιες ε, υποθέσεις με την Όλαφ. Ε, εγώ, επειδή είμαι εισηγήτρια για την εργασία τη Όλαφ, ε, πολύ θα με ενδιαφέρουν οι απαντήσει σα. Ούτω ή άλλω, σε μένα πρέπει να τι απευθύνετε. Πολύ καλό που μπορούμε να εργαστούμε προ την ίδια κατεύθυνση. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει επαρκέ προσωπικό σε όλε τι αρμόδιε υπηρεσίε. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι όμω θέμα μόνο δικό σα. Το θέμα είναι ότι η συνεργασία πρέπει να γίνει ούτως ώστε να υπάρχει σωστή ανταλλαγή πληροφοριών Κοιτάξτε, μπορεί να πει κανείς πολλά για την ανταλλαγή προφοριών, αλλά πρέπει να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή προφοριών για να καταλάβει η Ευρωπαϊκή Συγγελία πότε πρέπει να παρέμβει. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να είναι μόνιμη η ανταλλαγή προφοριών και εγγυημένη. Γιατί πρέπει να ξέρουμε σε κάθε φάση διαδικασίας τι μπορώ να κάνω εγώ. Τι μπορώ να κάνω τόσο ώστε να ανακτήσουμε τις ε, ε, απώλειες και να υπάρξουν συνέπειες όχι μόνο ποινικέ, αλλά και από πλευράς διοικητικών κυρώσεων. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε την ανάκτηση των ε, Η Όλαφ μπορεί να κάνει περισσότερα από πλευράς διοικητική, διοικητικής, να κάνει συγκεκριμένες συστάσεις. Εδώ λοιπόν ε, υπάρχει η αναγκαία συμπληρωματικότητα. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουν μέχρι το τέλο ποινική διαδικασία για να ξεκινήσουν οι διοικητικέ διαδικασίε. Πρέπει να υπάρχει αυτή η αναγκαία ανταλλαγή πληροφοριών για να υπάρχει η σωστή κατανομή εργασία μεταξύ αυτών των δύο θεσμών. Δεν είναι δυνατόν να πούμε, να πούμε ότι η Όλαφ απλώ συμβάλλει στην εργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία και όταν ολοκληρωθεί η εργασία της Εισαγγελίας τότε θα ε, ασχοληθεί και πάλι με την υπόθεση αυτή η Όλαφ. Όχι, πρέπει να υπάρχουν παράλληλε διαδικασίε και πρέπει να είναι εγγυημένε αυτέ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Α, όχι, ένα άλλο συνάδελφος. Ο κύριος Κον. Κάτι άλλο. Για την πείρα που έχετε με τι εθνικέ εισαγγελίε. Πείτε μας κάτι περισσότερο γι' αυτό παρακαλώ. Για το, γιατί η διεθνής και εθνική πείρα σα, ιδίως μετά την επανένωση της Γερμανίας, θα σας έκανε κατάλληλο για αυτή τη θέση. Όπως είπατε, υπήρξε μια ειδική κατάσταση στη δεκαετία του 90 στη Γερμανία, στα διάφορα ομοσπονδιακά κράτη. Γιατί δεν υπήρχαν ε, όλα όσα κατόπιν δημιουργήθηκαν. Αυτά που υπήρχαν δηλαδή στην ε, δυτική πλευρά. Χρειάστηκε λοιπόν να γίνουν σε ορισμένε εισαγγελίε ορισμένα πράγματα σε μία φάση, ενώ σε άλλε έγιναν πολύ αργότερα. Αυτό μου επέτρεψε πολύ νωρίς να συμμετάσχω σε προγράμματα ε, τεχνικής συνεργασίας και γι' αυτό πήγα στην ε, Λατινική Αμερική, στη Χιλή, την Παραγουάη και στο τέλος και στο Μεξικό για να ενημερώσω για το πώς πρέπει να δημιουργηθεί μία εισαγγελία όσον αφορά την ανεξαρτησία της και πώς τεχνικά πρέπει να οργανωθεί αυτή η εργασία. Και η πείρα που συνέλεξα είναι κάτι που ε, βοήθησε. Να σας το πω πολύ ανοιχτά, η πρώτη μου δραστηριότητα που ανέπτυξα στο 2000-2001, αυτές τις συμβουλές που έδωσα, θα ήταν πολύ διαφορετικές ε, αν τις έδινα τώρα. Γιατί εντωμεταξύ ε, είμαι 26 χρόνια σε αυτήν την υπηρεσία. Τώρα έχω περισσότερη πείρα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα μια εισαγγελία. Αυτά τα έμαθα και εγώ από την πείρα μου πώς μπορεί να κατανεμηθεί εργασία, πώς μπορεί να οργανωθεί συνεργασία, πώς μπορούμε να ε, εμψυχώνουμε τους συναδέλφους. Και ο τρόπος λειτουργίας μιας υπηρεσίας παίζει μεγάλο ρόλο στην επιτυχία της. Πρέπει βεβαίως να υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις. Εδώ, με τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχετε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. Τώρα πρέπει να εφαρμοστεί σε ένα βέβαια περίπλοκο περιβάλλον. Ευχαριστώ η κυρία Μακοβέη. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνεχίσω μετά την απάντηση που δώσατε στην πρώτη μου ερώτηση. Με μια δεύτερη Είπατε ότι δεν βιώσατε πολιτική πίεση. Οπότε, πώς θέλετε να αναλάβετε τη θέση του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα με 22 χώρες, όπου μερικές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης προσπαθήσουν να ασκήσουν πολιτική πίεση. Πώς θα το αντιμετωπίσετε. κυρία Μακοβέ. Σας ευχαριστώ πολύ και για αυτή την ερώτηση. Τι να σας πω. Η εργασία ενός εισαγγελέα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και η υπηρεσία του. Πρέπει να βασίζεται στις αρχές της νομιμότητας και να μην επηρεάζεται από άτομα. Για να μπορούμε να το εγγυθούμε αυτό, πρέπει να το αναλάβει, να αναλάβει την ευθύνη ο καθένας. Τώρα, ως απάντηση, ίσως να μην σας αρκεί. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο βέβαια να το κάνει κανείς αυτό. Η ανεξαρτησία ως έννοια δεν σημαίνει πως ούτως άλλως δεν θα υπάρχουν πολιτικές επιρροές. Δεν λειτουργεί ο εισαγγελέα εν κενό. Κάθε δραστηριότητά του μπορεί να έχει κάποια πολιτική σημασία και επιπτώσεις ανάλογα με πώς θα εξελιχθεί και θα καταλήξει. Αλλά ο εισαγγελέα πρέπει να το γνωρίζει αυτό, αλλά και επειδή το γνωρίζει, δεν θα πρέπει να ε, υποχωρήσει, αλλά να αντισταθεί αν υπάρχουν πιέσεις. Και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που υφίστανται τέτοιες πιέσεις παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά κάνουν σωστά τη δουλειά τους κάνουν όντως σωστά τη δουλειά τους. Και με το παράδειγμα τους και με τη δέσμευσή τους για το κράτος δικαίου αποδεικνύουν τι σημαίνει στην πράξη αυτή η ανεξαρτησία. Ευχαριστώ. Κανονικά θα έπρεπε να χειροκροτήσουμε εδώ. Παρακαλώ. Εσείς κύριε συνάδελφε. Άλλοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ρίτερ Καταρχήν ευχαριστούμε για τις γραπτές απαντήσεις που δώσατε στο ερωτηματολόγιο μας. Είναι αξιοθαύμαστο το βιογραφικό σας που έχει χρόνια σταδιοδρομία, πλούσια επαγγελματική πείρα. Είπατε ότι έχετε εμπειρία από συνεργασία με την ΟΛΑΦ. Και σίγουρα είναι προτεραιότητα η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με, με την ΟΛΑΦ. Δεν θα πρέπει όμως να δημιουργηθεί σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο στο μέλλον και επιβράδυση των ερευνών. Μπορείτε να μας καθησυχάσετε και να πείτε πώς βλέπετε αυτή τη συνεργασία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση και μετάδοση πληροφοριών. Η φιλελεύθερη πολιτική μου ομάδα ήταν υπέρ μια κεντρική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η τωρινή πρόταση είναι κάποια υβριδική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με κεντρικό φορέα αλλά και κάποια αποκεντρωμένα επίπεδα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότητα και ομαλή και γρήγορη διεξαγωγή των ερευνών. Πώ θα φροντίσετε να λειτουργήσει εύρυθμα αυτή η υβριδική δομή. Επίση, ε, πώ ε, θα προωθήσετε κάποιου διάβλου επικοινωνία για ομαλή και γρήγορη ε, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών και των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Ευχαριστώ. Συγκεκριμένα για το τελευταίο σας ερώτημα. Η συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει μόνο υπό τον όρο ότι υπάρχει ένα μηχανογραφικό σύστημα, σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο θα παρέχει τις, τις απαραίτητες πληροφορίες και για τον εντεταλμένο Ευρωπαίο Εισαγγελέα και για το σώμα. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ανταλλαγή προφοριών, προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει αυτή η, ανταλλαγή, η ζητούμενη ανταλλαγή προφοριών. Τώρα, αν καταλαβαίνετε, η, η, δομή λήψη αποφάσεων είναι περίπλοκη. Θεωρώ όμω ότι είναι η καλύτερη με απότερο στόχο να δημιουργηθεί μια, ομορφ... μια ομοιόμορφη διαδικασία λήψη αποφάσεων αντί να είχε, αντί να ε, είχε δημιουργηθεί εκ των προτέρων μια τέτοια ε, ε, δομή. γιατί θα απαιτούνταν ένα επίπεδο εναρμόνισης το οποίο θα ήταν και ανέφικτο αν θέλετε τη, τη γνώμη μου. Πρέπει πραγματικά να, να ληφθούν υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες των εθνικών συστημάτων, των δικαιικών συστημάτων, ε, ώστε να υπάρχει ε, αποτελεσματική ε, ποινική δίωξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια κάθετη προσέγγιση, όσο ενδιαφέρουσα και αν μπορεί να φαινόταν, στις τρέχουσες συνθήκες δεν θα ήταν ε, η ιδανικότερη λύση. Ακριβώς αυτή, αυτός ο υβριδικός χαρακτήρας μας επιτρέπει ε, να αξιοποιήσουμε τα καλύτερα στοιχεία και του ευρωπαϊκού και του εθνικού επίπεδου για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων μας. Για τη συνεργασία με τον ε, Όλαφ, το είπα και νωρίτερα, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχή ροή πληροφοριών. Να μην μα ενημερώνει δηλαδή ο Όλαφ μόνο στην αρχή τη διερέυνησης μια υπόθεση και να τελειώνει εκεί ο ρόλος του. Να υπάρχει συνεχώς και αδιαλείπτως μια ροή νέων στοιχείων και πληροφοριών. Ευχαριστώ πολύ. Viter urat a meghallgatáson. Két kérdést szeretnék föltenni. Az egyik, hogy továbbra is több tagállam nem csak... No translation. No translation? Okay, then I continue in English. Αν δεν υπάρχει διερμηνία, να μιλήσω αγγλικά. Έχω δύο ερωτήσεις. Ε, έχουμε κάποιες χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει ακόμη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι σκοπεύετε να κάνετε αν σε μια έρευνα διασυνοριακού εγκλήματος ανακαλύψατε ότι κάποια τμήματα της έρευνας πρέπει να γίνουν στα κράτη-μέλη που δεν προσχώρησαν ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για διενέργεια ερευνών. Πώς θα εξασφαλίσετε σωστή διερεύνηση αυτών των διασυνοριακών εγκλημάτων, ιδιαίτερα όταν κάποια τμήματα τη έρευνα θα πρέπει να γίνουν σε χώρε που δεν έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ένα άλλο θέμα που έχει συζητηθεί ιδιαίτερω. Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΟΛΑΦ και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την εμπειρία μα με την ΟΛΑΦ γνωρίζουμε ότι μερικέ φορέ το πρόβλημα είναι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και τη ΟΛΑΦ ή των άλλων ευρωπαϊκών φορέων. Ίσως το ίδιο πρόβλημα ανακύψει και στις σχέσεις ε, η ανταλλαγή ε, πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι θα κάνετε αν κράτη-μέλη συστηματικά σα αρνούνται παροχή πληροφοριών για συγκεκριμένο έγκλημα που ερευνάτε. Αναφέρεστε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Προφανώς αν δεν έχει τις κατάλληλε πληροφορίε στη διάθεσή της, δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι πληροφορίε, λοιπόν από τα κράτη-μέλη, από, του, από τους οργανισμούς, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άλλωστε δεν θα είχε και υποθέσει να χειριστεί. Άρα πρέπει τα πράγματα να διαμορφωθούν και να εφαρμοστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι λειτουργικά και αποτελεσματικά. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει να δημιουργηθούν και οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις ε, να μπορούν να παραλαμβάνονται πληροφορίες και από τρίτα πρόσωπα. Από πληροφοριοδότες, για παράδειγμα, καταγγέλλοντες. Να υπάρχει δηλαδή και ένας άλλος εναλλακτικός, αν θέλετε, διάβλος ε, ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Γιατί ξέρετε ότι άλλωστε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να δεν παραλαμβάνει μόνο πληροφορίες, αλλά μπορεί και να ζητεί, να αναζητεί η ίδια τι ε, πληροφορίε που χρειάζεται όσον αφορά τις διασυνοριακές δραστηριότητες με τα κράτη που δεν συμμετέχουν. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που μας παρέχει η Eurojust. Γιατί εκεί θα υπάρχει αρμοδιότητα της Eurojust, όχι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία. Μέσω κοινών ομάδων διερεύνησης, λοιπόν, στις οποίες θα συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μαζί με τα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νομίζω ότι αυτό θα είναι η καλύτερη δυνατότητα συντονισμού των ερευνών και να αποφευχθεί στο βαθμό και στο μέτρο του δυνατού ο κατακαιρματισμός των προσπαθειών για την υπεράσπιση των οικονομικών ε, συμφερόντων της Ένωσης. Ο κύριος Σομαρζέ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Ρίτερ, έχω δύο ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Από τη μακροχρόνια πήρα και στα διαδρομία σας Αντιμετωπίσατε κάποια πολιτικο-οικονομικά θέματα, υποθέσεις διαπλοκής και χρειάστηκε να διώξετε πολιτικούς ερετούς. Ε, ε, εκφράστε ανησυχίες γιατί αναγνωρίσετε το ενδεχόμενο άσκησης πολιτικής πίεσης ε, στους ε, εισαγγελείς στα κράτη-μέλη. Μάλιστα, η συνάδελφος η κυρία Κοβέτζη έχει υποστεί κριτική και επίθεση από την κυβέρνηση της χώρας της. Ποια είναι η γνώμη σας για την κατάσταση αυτή. Αν θέλετε φυσικά να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Μπορώ να σας απαντήσω σύντομα. Απάντηση στο πρώτο ε, σας ερώτημα. Αν, είχ, αν χειρίστηκα υποθέσεις κατά ερετών και αν μου ασκήθηκε πολιτική πίεση. Ναι, χειρίστηκα τι υποθέσει, πολιτική πίεση δεν δέχτηκα. Δεν μπορώ να ισχυριστώ κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά την ε, κατάσταση που επικρατεί σε άλλες χώρες και ποια είναι η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν οι συνοψήφοι μου. Εγώ μπορώ να σας πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή να ανήκω σε αυτόν τον ε, κατάλογο υποψηφίων στον οποίο ανήκει και η κυρία Κοβέση, την οποία θαυμάζω για το θάρρος της και για όλα όσα έχει κάνει. Και νομίζω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους δύο συνυψοψηφίους μου, μπορώ να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή που ανήκω σε αυτή την τριάδα των επικρατέστερων υποψηφίων. Το EFDD δεν θέλει το λόγο, Κυρία Πιτέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στην ερώτηση του κυρίου Γιάβορ. Στο γεγονός δηλαδή ότι δεν έχουν προσχωρήσει, δεν συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη με την σύσταση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Οπότε θα είναι ενδιαφέροντα τα θέματα συνεργασίας με χώρες που δεν στηρίζουν αυτό το σχέδιο, αυτή την πρωτοβουλία σύσταση Ευρωπαϊκής Αγγελικής Αρχής. Και οι χώρες που δεν, δεν συμφωνούν με αυτό το σχέδιο, δεν το έχουν εγκρίνει, σε μεγάλο βαθμό θεωρούν ότι η δημιουργία Ευρωπαϊκής Αγγελίας αφαιρεί από τις εθνικές εισαγγελίες την ανεξαρτησία τους ή πλήττει την ανεξαρτησία των εθνικών εισαγγελιών. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει απειλή για την ανεξαρτησία των εθνικών εισαγγελέων. Πώς θα διασκεδάζετε τέτοιες ανησυχίες που έχουν εκδηλώσει οι χώρες μέλη. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής εισαγγελία, στην οποία κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία των λειτουργών της, θα μπορούσε να περιορίσει την ανεξαρτησία των εθνικών εισαγγελικών αρχών. Υπάρχουν σαφώς οριοθετημένοι τομείς, εντός των οποίων θα δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στους τομείς αυτής εξασφαλίζεται με τέτοιον τρόπο μέσω του κανονισμού η ανεξαρτησία της αλλά και μέσω της ε, υποχρέωσης λογοδοσίας σε εσάς Νομίζω ότι πραγματικά κανένα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι περιορίζεται η ανεξαρτησία των εθνικών εισαγγελέων από το έργο τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να, να κατανοήσω ούτε να παρακολουθήσω ένα τέτοιο συλλογισμό. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Επιτροπή ε, Ελέγχου του Προπολογισμού, ε, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σα. Ήταν τιμή μα που σα γνωρίσαμε. Ευχαριστώ θερμά του ευρωβουλευτέ για τι ερωτήσει και ευχαριστώ και τον κύριο Ρίτερ για τη συμμετοχή στην ακρόαση αυτή. Μάλιστα μετά την ακρόαση θα γίνει μια πλήρης αξιολόγηση των ακροάσεων με τους τρεις υποψηφίους και θα ενημερώσω πλήρως τα μέλη για το πώς θα γίνουν οι αξιολογήσει των δύο επιτροπών, αφού ολοκληρώσουμε όμω και τις τρεις ακροάσεις. Μετά από έτοιμα του Πρόεδρου Ταϊγιάννη έστειλα απαντητική επιστολή και αφού ολοκληρώσουμε τις αξιολογήσεις, θα στείλω και δεύτερη επιστολή στον Πρόεδρο Ταγιάννη με το αποτέλεσμα των, ε, αξιολογήσεων και τη γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Έρχεται και ο δεύτερος μας υποψήφιος, βρίσκεται καθοδόν, δεν θα έχουμε μεγάλη καθυστέρηση, φαντάζομαι σε λιγότερο από ένα λεπτό θα είναι στην αίθουσα. Colleagues. Just again, the, the, the point I was making about movement and so on, thank you. Appreciate it, thank you. So, θα ήθελα παρακαλώ να καθίσετε και να δείξουμε σεβασμό προς καλεσμένους μας, τους υποψηφίους. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Ζαν Φρανσουά Μπονέχ, το δεύτερο υποψήφιο να επαναλάβω αυτά που είπα και για τον πρώτο υποψήφιο. Γιατί ο κύριος Μπονέρ πρώτη φορά έρχεται και δεν ξέρει τη διαδικασία. Θα ακούσουμε την εισαγωγική τομιλία που δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 7 λεπτά και θα ακολουθήσει γύρω σε ερωταπαντήσεων. 63 λεπτά θα κρατήσει, 14 ερωτήσεις θα θέσουν μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και 7 της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Ε, θα έχουμε ερωτήσεις που θα κρατούν ένα λεπτό και απαντήσεις δύο λεπτά θα είμαστε πολύ αυστηροί με την τήρηση του χρόνου ομιλία. Αλλιώ δεν θα μείνει χρόνο για την τρίτη υποψήφια. Γι' αυτό λοιπόν θα τηρήσουμε πολύ πιστά το χρόνο ομιλία, οπότε το μάτι σα και στο χρονόμετρο. Έχουμε διερμηνία, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μητρική σα γλώσσα, αλλά προσοχή να μην μιλάτε πολύ γρήγορα για να σα προλαβαίνουν και διερμηνεί. Χωρί άλλη καθυστέρηση, να δώσω το λόγο στον κύριο Μπονέρ για να μα κάνει την παρουσίαση που θα κρατήσει το πολύ 7 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα να εκφράσω μια σκέψη αυτή τη στιγμή για έναν από τους πρώην Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Κλάους Χένς, που πριν από 23 χρόνια, το 1996, ανέφερε για πρώτη φορά την ιδέα της σύστασης μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έρχομαι σήμερα εδώ ενώπιόν σας με μια διπλή πύρα, την πύρα του Ευρωπαίου Δικαστή και την πύρα του πεπειραμένου εισαγγελέα. Ήμουν Ευρωπαίος Δικαστής ε, με 20 ετή σταδιοδρομία που αφιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή Δικαστική Συνεργασία, επιχειρησιακή συνεργασία. Αλλά ε, έχω και άλλη εμπειρία. Συνέβαλα στο Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα μια και δύο φορές είχα την τιμή να συμμετέχω ή να πρωτοστατώ στη δημιουργία δύο βασικών νομικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Δικαστικής Συνεργασίας. Τη δημιουργία της θέσης του Ευρωπαίου Δικαστή Συνδέσμου και την δημιουργία της Eurojust, της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας. Ήμουν και ο Γάλλος εκπρόσωπος. Είμαι πεπισμένο και μεγάλος τη Ευρωπαϊκής Ένωση. 32 χρόνια είχα σταδιοδρομία στην εισαγγελία και από αυτά τα 32 χρόνια 14 αφιερώθηκαν στην καταπολέμηση του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού εγκλήματος ε, κάθε μορφής. Γιατί είχαμε κυρίως ε, απάτες στα μέσα πληρωμής και στη συνέχεια όταν άλλαξαν οι αρμοδιότητε, ανέλαβα πολύ πιο περίπλοκες υποθέσεις, απάτες στο ΦΠΑ, νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διαφθορά, οργανωμένο έγκλημα, κατάχρηση δημόσιων αγαθών και ούτω καθεξής. Δέκα χρόνια της σταδιοδρομίας μου αφιερώθηκαν και συνεχίζονται να αφιερώνονται σε, ε, στη θέση μου ε, επικεφαλής ε, Γενικός Εγγελέας και σήμερα, μετά από μια τοπική θητεία, ε, είμαι επικεφαλής Γενικός Εισαγγελέας ε, σε μια περιφερειακή εισαγγελία. Και είμαι τώρα στη διάθεσή σας και μπορώ να υπηρετήσω και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ε, είχα επαφή με επαγγελματίε από πολύ διαφορετικούς νομικούς και δικαστικούς ορίζοντες και τους είδα να εξελίσσονται ε, μαζί μου σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον. Και θα ήθελα να αξιοποιήσω όλες τις πιθανές συνέργειες και να ψυχώσω όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να συστήσουμε μια αλληλέγγυα ομάδα ενωμένη που θα εργάζεται σε ένα ε, νυφάλιο κλίμα. Και το σύνθημά μου θα είναι ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και εννοείται και η ιδεοντολογία. Και γι' αυτό θα χρειαστεί συνένεση, διπλωματικότητα, αλλά πάνω απ' όλα πυγμή και αποφασιστικότητα, όπως χρειάζεται στο πρόσωπο ενός επικεφαλής ε, εισαγγελική αρχής. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει από την αρχή να αντιμετωπίσει τρεις βασικές προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χρειάζεται πρώτα απ' όλα αξιοπιστία ως νέο ευρωπαϊκό σώμα, ω νέο Ευρωπαϊκό φορέας και εν μέσω των εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστικών αρχών ε, φορέων και ε, μονάδων επιβολής του νόμου θα πρέπει να τοποθετηθεί. Και η βασική ε, αρμοδιότητα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα είναι να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο δρόμο της απόκτησης νομιμοποίησης που θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση της αξιοπιστίας που χρειάζεται. Εν συνεχεία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να πείσει. Να πείσει τις 22 χώρες μέλη που συμμετέχουν σε αυτή τη δομή να συνεργαστούν μαζί της και να μεταβιβάζουν τις υποθέσεις της αρμοδιότητάς τους. Επίσης, θα πρέπει να πείσει και τις έξι αναπομείνασες χώρες που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να βοηθήσουν την αρχή αυτή όπου είναι αναγκαίο και όπου χρειάζεται όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης θα πρέπει να πιστούν. Και ενώ κυρίω την ΟΛΑΒ, την Eurojust και την Ευρωπόλ. Και ο κύριος σύνδεσμος μεταξύ των τεσσάρων φορέων, γιατί περιλαμβάνω εδώ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα πρέπει να είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Τουλάχιστον θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οφείλει να δώσει και νέες προοπτικές για την Ευρώπη. Και από τότε που τη γνωρίζουμε, τα δημοκρατικά θεμέλια αμφισβητούνται και τίθενται ένα αμφιβόλο σε πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με την αποτελεσματική καταπολέμηση ε, των ε, οικονομικών εγκλημάτων και με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και καταπολεμώντας κάθε μορφή εγκληματικότητας, συμπεριλαμβανομένης και της διαφθοράς, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα εμφανιστεί σίγουρα ως το νέο μέσο, το νέο εργαλείο της εμπιστοσύνης στη δημοκρατία. Τέλος κυρίες και κύριοι. Πέρασα πριν από λίγο την Μπασαρέλα Κόνραντ Αντενάουερ. Θα ήθελα λοιπόν να θυμηθούμε τον ε, καγκελάριο Κόνραντ Αντενάουερ που κάποτε είπε ότι η παγκόσμια ιστορία είναι το άθροισμα όλων όσων θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί κατά την ε, δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας έχουμε ενώπιον μας μια τεράστια πρόκληση. Αλλά παράλληλα ε, είμαστε και ενώπιον μιας μεγάλης να δημιουργήσουμε ένα νέο μέσο δημιουργίας ε, δημοκρατικής εμπιστοσύνης της κοινή γνώμης. Σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Το οφείλουμε στους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, uh, Monsieur Bonner. We now... Ευχαριστώ κύριε Bonner. Και τώρα ερωτήσεις. Λοιπόν, πρώτα το ΕΛΚ. Ο κύριος ε, Έγκο για ένα λεπτό. Ο κύριος Εγγέλ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπονέα έχετε το ίδιο επώνυμο με τον ε, γυμνασιάρχη μου. Τον παλιό γυμνασιάρχη μου. Άρα σας αισθάνομαι κοντά μου. Κοιτάξτε, υπάρχουν και κάποια κρατημέλη που δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ίσως λοιπόν να έχουν ε, καλούς λόγους. Δεν είναι μόνο θεωρητικοί λόγοι δικαστικής και εθνικής ανεξαρτησίας. Αν λοιπόν αναλάβετε το αξίωμα, πώς θεωρείτε ότι το κύρος του αξιώματός σας θα μπορούσε να βοηθήσει ούτως ώστε να πείσουμε όσους δεν συμμετέχουν να συμμετάσχουν. Και πώς το κύρος σας θα μπορούσε να βοηθήσει ούτως ώστε να αποφύγουμε εξαρτίες δυσφήμισης όπως αυτές που γίνονται από πλευρά των ρουμανικών αρχών κατά τη συνυποψηφία σας από τη χώρα αυτή. Μια που θέλετε να μιλήσουμε για ε, απευκταία ενδεχόμενα. Ε, ναι, για το πρώτο τμήμα της ερώτησής σας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει. Πρέπει να αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να καταπολεμήσει αποτελεσματικά κάθε παράβαση που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Αυτή είναι η, ουσία των αρμοδιοτήτων της. Ε, βέβαια δεν ξεχνάω τα άλλα δικήματα, η διαφθορά, η κατάχρηση δημοσίων αγαθών ή η οργανωμένη εγκληματικότητα βεβαίως ε, είναι σημαντικά, αλλά πρέπει να συνδέονται με τις παραβάσεις ε, κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Αυτή είναι η πρώτη αρμοδιότητα και αποδεικνύεται ότι μπορεί αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει αυτές τις παραβάσεις, αυτά τα δικήματα, ε, δίνοντας συγκεκριμένα αποδείξεις και έναντι των έξι άλλων κρατών μελών ότι μπορεί να λειτουργήσει, ίσως θα μπορούσε να αλλάξει τη στάση τους. Τώρα για το δεύτερο θέμα. Θα έλεγα ότι έχουμε μια κατάσταση που πρέπει όντως ε, να αντιμετωπίσει ο επικεφαλής της εισαγγελία. Νομίζω ότι η σωστή συμπεριφορά θα πρέπει να είναι για τον ε, Ευρωπαίο Εισαγγελέα να βασιστούμε στα κείμενα, στον κανονισμό δηλαδή. Καθορίζει την αποστολή μας, το νομικό πλαίσιο, πρέπει οπωσδήποτε να τα σεβαστούμε αυτά, να αποδείξουμε ότι μέσω της εφαρμογής των κειμένων η εισαγγελία είναι όντως ε, ανεξάρτητος θεσμός και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι ακριβώς αυτή που πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να σεβαστεί αυτή την ανεξαρτησία, ούτω ώστε και τα άλλα κρατημέλη και άλλοι θεσμοί να επηρεαστούν και να ε, λειτουργήσουν και αυτοί ανεξάρτητα. Αναφέρατε ορισμένα, υπάρχουν και άλλα. Για τους σοσιαλιστές. Η κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ κύριε Μπονέα έχοντας κατά νου τα διαφορετικά ε, συστήματα δικαιοσύνης που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Μπορείτε να μας εξηγήσετε μήπως εσείς ε, θα μπορέσετε να συμμορφωθείτε ή συμμορφώνεστε, εν πάση περιπτώσει, εκπληρώνετε όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρει στο άρθρο 14 ο κανονισμός. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ότι πρέπει να είναι αδιαμφισβήτητη η ανεξαρτησία σας και ότι έχετε ε, και τα προσόντα για να διοριστείτε στην υψηλότερη δυνατή θέση εισαγγελέα στη χώρα σας. Σας ευχαριστώ. Ανεξαρτησία και προϋποθέσεις. Να ξεκινήσω με το τελευταίο. Ως προϋποθέσεις, όπως είπα και πριν από λίγα λεπτά, εγώ έχω περάσει από όλες τις θέσεις της εισαγγελία στη Γαλλία. Από ε, τις χαμηλότερες έως τις υψηλότερες θέσεις έχω αξιοποιήσει όλα τα μέσα που παρέχει ο νόμος ε, στην στη Γαλλική Εισαγγελία για να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην υψηλότερη δυνατή θέση που μπορεί να φτάσει ένας εισαγγελέα στην Γαλλία. Ήμουν λοιπόν νέος εισαγγελέα, στη συνέχεια ε, ε, ανέβηκα στην ιεραρχία σε συνεργασία και με, ευρωπαϊκές, με άλλες ευρωπαϊκές εισαγγελίες και τώρα πλέον είμαι ο πρεσβύτερος εισαγγελέα και νομίζω ότι εκπληρώνω όλες τις προϋποθέσεις που περιγράφει ο κανονισμός. Όσον αφορά την ανεξαρτησία, Κάποιες φορές λέγεται ότι το γαλλικό σύστημα στο παρελθόν ήταν πολύ ιεραρχικό. Κάτι που σήμαινε ότι στο παρελθόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορούσε να δώσει οδηγίες στον ε, Γενικό Εισαγγελέα. Αυτό πλέον έχει αλλάξει εδώ και έξι χρόνια. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν μπορεί πλέον να δίνει οδηγίες στον ε, Γενικό Εισαγγελέα σε συγκεκριμένε υποθέσεις Και αυτό ε, αποτελεί μια μεγάλη μεταστροφή όσον αφορά την κουλτούρα μα ω ε, Γενικών Εισαγγελέων στην Γαλλία, πρέπει να σα πω. Και βλέπω ότι και οι νέοι εισαγγελεί που αναλαμβάνουν τώρα τα καθήκοντά του έχουν πραγματικά αυτό κατά νου όταν εκπληρώνουν τα καθήκοντά του. Ευχαριστώ. Η Χέλγα Στίβενς για το ECR έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Μπονέρ. Στις γραπτές σας απαντήσεις αναφερθήκατε στην περίπλοκη σχέση ε, που θα έχουν οι εθνικές εισαγγελίες με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πείτε μας λίγα περισσότερα. Πώς ακριβώς θα καταφέρετε εσείς να επιτελείτε δεν υπήρχε διερμηνία ε, από ό,τι ακούμε, οπότε η κυρία Στίβενς μάλλον θα ξεκινήσει. Στα ελληνικά υπήρχε διερμηνία, δεν υπήρχε διερμηνία στα αγγλικά όμως από ό,τι φαίνεται. Ξαναξεκινώ λοιπόν. Κύριε Μπονέρ. Στις γραπτές σας απαντήσεις αναφέρεστε στην περίπλοκη σχέση που θα έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τις μη συμμετέχουσες χώρες. Μήπως μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες στοιχεία. Ποια μέσα θα έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη διάθεσή της ώστε να χειρίζεται διασυνοριακές υποθέσεις οι οποίες, στις οποίες εμπλέκονται και οι μη συμμετέχουσες χώρες. Ίσως Υπάρχουν και πολιτικοί λόγοι για κάποιες χώρες για το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν, οπότε αντιστοιχώ ενδέχεται να ασκηθεί και πολιτική πίεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Χέλγα Ευχαριστώ και συγγνώμη για τη διακοπή αυτή. Κύριε Μπονέχ. Eh, eh, Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι θέτεται αυτό το ζήτημα και το ότι θα πρέπει να βλέπω ε, ότι ε, δείχνετε και τις πολλές σας ε, γλωσσικές ικανότητες. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει πράγματι ένα τμήμα της ε, νομοθεσίας που προβλέπει σήμερα ότι σε κάθε περίπτωση οι χώρες που οι μη συμμετέχουσες θα συνδέονται στα, με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη μέσω της αρχής της ειλικρίνειας της συνεργασίας. Έχουμε λοιπόν του συσχετισμού τη εισαγγελία στα κρατημέλη που θα είναι σε θέση να θέσουν στη διάθεσή του τα μέσα που θα έχει η εισαγγελία συμπεριλαμβάνων των ενταλμάτων στο σύνολο της επικρατείας και προς τα κράτη που δεν θα συμμετέχουν. Τώρα το ερώτημα είναι λίγο πιο περίπλοκο ή στο βαθμό που γνωρίζω ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει να διερευνήσει κατά πόσον θα έχουμε συμπληρωματικό μέσο που θα συνδέει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τα μη συμμετέχοντα κράτη. Αυτό το ερώτημα είναι εκρεμές και άπτεται εν πάση περιπτώσει νομικών ζητημάτων δεν γνωρίζω αν είναι νομοτεχνικά τα ζητήματα και οπωσδήποτε θα ήταν ένα από, μία από τις πρώτες προτεραιότητές μου, δηλαδή να εξασφαλίσω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι σε θέση να συνεργάζεται απολύτως καλά με τα κράτη αυτά μέλη. Και θυμίζω ότι στην περίπτωση που θα χρειαζόταν θα καθότι η Eurojust καλύπτει το σύνολο των 28 σήμερα των μελών, αυτό θα μας βοηθούσε να υπερβούμε το οποιοδήποτε νομικό κόλλημα ή εμπόδιο. Η κυρία Ζουλή για τους ε, πρασίνους ε, όχι, ζητώ συγγνώμη Εύα, λέει ο Πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη. But, um, for the Audi group, Natalie ε, η Νάταλη για το, για το Aldi. La question sera posée en français et ε, euh, de la question de, de ma collègue Elga Stevens, vous avez évoqué... Μιλήσατε στην παρουσίασή σας για το σύνολο των μέσων που θα έχουμε στη, στη διάθεσή μας και αναφέρομαι εγώ στη σχέση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και των κρατών μελών ακριβώς που δεν συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην εισαγγελία. Πώς φαντάζεστε ότι οι εθνικοί ανταποκριτές της Eurojust, της Eurojust με συγχωρείτε, θα συνεργάζονται, πώς δηλαδή θα εργάζονται ώστε τα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν δεν θα παρεμποδίζουν εντός εισαγωγικών το τη δουλειά της αγγελίας. Και δεύτερο ερώτημα, ταχύτατα. Κατά την προετοιμασία του κανονισμού, ένα από τα ερωτήματα, μία από τις απορίες θα ήταν ότι ακριβώς δεν θα ήταν ενδεχομένως επαρκώς ευρωπαϊκή εστίαση. Δηλαδή, ποια μέτρα θα λαμβάνατε υπόψη σας, θα λαμβάνατε, για να είναι πιο αποτελεσματική η εργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κοιτάξτε, να σας απαντήσω. Για την Eurojust μιλούμε για ένα στοιχείο που θα είναι ουσιοδέστατο, γιατί θα είναι ακριβώς ο σχετισμός μεταξύ της εισαγγελίας, εισαγγελίας και της Eurojust. Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή το βαθμό κάλυψης της Eurojust που είναι το σύνολο του ευρωπαϊκού εδάφους και ακόμα παραπέρα διότι έχουμε υπογράψει, Eurojust έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με τρίτες χώρες. Έχουμε δικαστικούς επαφής, Νορβηγούς, Αμερικανούς, αυτούς που υπόκεινται στη συμφωνία συνεργασίας και μια δυνατότητα αποσύνδεσης, αν θέλετε, με την ακτίνα δράσεως της Eurojust. Από εκεί και πέρα φυσικά θα πρέπει κανείς να αναπτύξει σχέσεις εργασίας πάρα πολύ με τους υπευθύνους αυτούς επαφής, ώστε οι άξονες αυτής της συνεργασίας να αναπτυχθούν και να τοποθετηθούν κανόνες επικοινωνίας ασφαλής και χωρίς επικαλύψεις. Ώστε η επικοινωνία να τρέχει ομαλά και ταχαίως Όπω το κάνει σήμερα η Eurojust όταν υπάρχουν συναντήσεις συντονισμού για μια ανακριτική ερευνητική συνεργασία. Τώρα για του εισαγγελεί του αποσπασμένου. Αυτό είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαστε από την αρχή. Σύμφωνα με την νομοθεσία θα γνωρίζετε ότι είναι δυνατόν να έχουμε ε, Ευρωπαίο εισαγγελέα κάθε αυτό, δηλαδή μόνο με αυτή την δικότητα και αποσπασμένο επομένως με τις δύο εντολές αν θέλετε. Εκεί χρειάζεται και πάλι στενή συνεργασία και συζήτηση με τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να διατηρήσουν αυτήν την δυνατότητα απόσπασης. Γιατί ίσως αυτό να είναι μια πηγή περιπλοκών ή εν πάση περιπτώσει λεπτομερών διευθετήσεων που θα πρέπει να αναλάβει εν τέλει ο εισαγγελέα. Σα ευχαριστώ κυρία Τζολή τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Γενικό Εισαγγελέα ε, σχετικά με τη συνεργασία για τρομοκρατικό επεισόδια και περιβαλλοντικά εγκλήματα. Επίσης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι για το όραμά σας της ανεξαρτησίας, όπως ε, όλοι ήταν σε θέση να το σημειώσουν στην, στην υπόθεση Μπεναλά, κατά πόσον έχετε ξεκινήσει έρευνες ε, επί τη βάση των πορισμάτων του, των Panama Papers και την βιομηχανία ξεπλήματος στην οποία βασιζόταν μια σειρά από τραπεζικά ιδρύματα. Αν αυτά ε, εμπίπτουν στο δίκτυό σας, σας ευχαριστώ κυρία μου για την διεύρυνση των της του ε, είναι το, το κεντρικό ερώτημα το οποίο την απάντηση περιμένουν όλοι. Κοιτάξτε, στα γονίδια θα έλεγα της Εβραϊκής Αγγελίας όταν θα έχει απογειωθεί, για να το πω έτσι μεταφορικά, και θα έχει αποκτήσει ένα επαρκές ύψος, υπό το 86 άρθρο της Λισαβόνας θα πρέπει να αναπτύξει τη δραστηριότητά του περαιτέρω. Αλλά Α είμαστε επιφυλακτικοί. Όπως λένε οι Άγγλοι φίλοι μας, οι Αγγλόφωνοι εν πάση περιπτώσει, step by step. Θα πρέπει να μπορεί και να διατηρήσει το αεροσκάφος τη Αγγελία το ύψος που θα έχει ανακτήσει. Θα πρέπει δηλαδή τα προηγούμενα που θα απαιτούνται να τα έχουμε καλέψει προ... προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε περαιτέρω δραστηριότητα η συνεργασία. Ίσως τα κρούσματα τρομοκρατίας, ίσως τα οικολογικά εγκλήματα, τα περιβαλλοντικά εγκλήματα γιατί υφίστανται, να είναι μια δυνατή περιοχή, ένα δυνατό πεδίο. Πάντως όλα τα σοβαρά εγκλήματα, τα διασυνοριακά θεωρητικά εμπίπτουν. Και επομένως μιλούμε για ένα ευρύτατο πεδίο, δεν αποκλείω καμία από τις περιοχές αυτές. Για την άλλη παρατήρησή σας για, ε, για τα θέματα ανεξαρτησίας και τα Panama Papers, στα έγγραφά μας έχουμε ερευνήσει λεπτομερέστατα προς όλες τις δεν θα αναφερθώ τώρα σε, τρέχους, σε τρέχοντες φακέλους, γνωρίζουμε ότι σήμερα είναι η αρμοδιότητα του Γενικού Εισαγγελέα και πολύ λιγότερο των Υπουργείων Δικαιοσύνης να δούμε τη δουλειά των αποσπασμένων εισαγγελέων που δουλεύουν για το γραφείο μας και αυτό οπωσδήποτε θα είναι αρμοδιότητα του επικεφαλή τη υπηρεσία αυτή. Η κυρία Μετσόλα. Um, Λυπάμαι πολύ που κάνω τέτοια λάθη. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη από την ΚΟΕ. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω καμία απορία για την ανεξαρτησία της αγγελίας. Έχω όμως Έντονε αμφιβελίες για την ανεξαρτησία των εθνικών εισαγγελιών στα κράτη-μέλη. Δηλαδή η θετική τοποθέτησή σα για την θεωρητική ανεξαρτησία, ανεξαρτησία της γαλλικής δικαιοσύνης εμένα μου γύρει σοβαρά ερωτηματικά. Εγώ ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποια είναι τα συγκεκριμένα μέσα που θα έχετε στη διάθεσή σας για να αντιμετωπίσετε τα ελλείμματα ακριβώς ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης σε συγκεκριμένα κρατημέλη. Και δεν μου φτάνει να ακούσω λόγια όπως πρέπει να ε, ε, ε, ασκήσουμε πειθό, να δημιουργήσουμε ερθετικό κλίμα, να είμαστε να μιλούμε πολλές γλώσσες. Δεν, δεν μου αρκούν αυτά. Δεν μου αρκεί να έχουμε διπλωματική μύτη και πνεύμα. Γιατί από μια πραγματική εισαγγελία δεν περιμένω καμία διπλωματία, να σας πω. Ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι ο, Ευρωπα... ο Ευρωπαίος Εισαγγελίας θα χρειαστεί πολύ και όχι καθόλου διπλωματία. Όμως, για το θέμα της ανεξαρτησίας έχετε δίκιο είναι κάτι που είναι απαραίτητο και δεν είναι κάτι που μπορούμε να το διατάσουμε, να το επιθυμούμε και άρα να υπάρχει. Στη Γαλλία, στη Γαλλία με συγχωρείτε, έχει αλλάξει η προσέγγιση των πραγμάτων αυτών και εγώ το γνωρίζω διότι έχω βιώσει την, το πεδίο αυτό, την περιοχή αυτή. Εγώ αν είχα ως καθήκον Θα, έχω προσεχώς, ε, θα είμαι ε, προσεχώς 58 ετών με 7 έντια εντολή θα έφτανα στα 65, δεν θα είχα τίποτα να περιμένω από την Γαλλική Εισαγγελία. Από τη Γαλλική Δικαστική Αρχή. Δεν θα είχα καμία εξάρτηση επομένω. Τώρα για τα μέσα, και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, θα εξαρτάται από το Γενικό Εισαγγελία σε καθημερινό επίπεδο από τις επιμέρους εισαγγελίε και από τους αποσπασμένους εισαγγελίες, που θα είναι το μόνιμο θερμόμετρο αν θέλετε του πώς θα λειτουργεί το όλο σύστημα να εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν αποκλήσεις ή ελλείμματα ανεξαρτησίας και τότε θα πρέπει ο επικεφαλής της εισαγγελίας όπως το είδα και στην εμπειρία μου από την Eurojust όταν έχουμε δυσλειτουργίες σε επίπεδο κρατου μέλου, κακή συνεργασία, ελλειπή συνεργασία, στην ετήσια έκθεση τότε στην Eurojust, το αναφέραμε και αυτό είχε συνέπειε. είχε αντίκτυπο. Και η πρώτη μου υποχρέωση είναι απέναντί σα, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί ενώπιόν σας θα πρέπει να υποβάλλω τέτοια ζητήματα δείχνοντα το δάχτυλο ενδεχομένω αν χρειαστεί το ένα ή το άλλο κράτο μέλο. Η κυρία Μετσόλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πέρα από τα όσα μας είπατε ήδη, μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερο όσον αφορά τις εμπειρίες σας σε υποθέσεις ε, μεγάλης προβολής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, και στο κοινό. Γνωρίζουμε ότι ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα πρέπει να χειριστεί κάποιες από τις ε, πιο πολιτικά φορτισμένες υποθέσεις. Είδαμε περιπτώσεις ε, στην Ευρώπη όπου οι αρχές επιβολής του νόμου αρνήθηκαν να αναλάβουν δράση, ε, πόσο μάλλον να διώξουν σαφείς σαφή εγκλήματα. Τι θα κάνετε με τα κράτη-μέλη που δεν συνεργάζονται και μπορείτε να μας δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα όπου ε, οργανωμένες εγκληματικές, όπου εγκληματικές οργανώσεις προσπάθησαν να ε, εξαπατήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ε, καταχραστούν πόρους. Όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπορώ να σας πω ότι στην προηγούμενη θέση ως επικεφαλής εισαγγελέα είχα μια εμπειρία που έπρεπε να διώξω έναν ανώτατο αξιωματούχο με τον οποίον ε, ε, ήμουν αναγκασμένος να συνεργάζομαι τακτικά ε, μία φορά την εβδομάδα στο πλαίσιο της νομαρχίας μας, της Prefecture. Και αυτός ο ανώτατος αξιωματούχος έπρεπε να διωχθεί για κατάχρηση, υπεξαίρεση. Και όχι από τη δική μου πλευρά, αλλά από άλλε ε, ε, πλευρές έφτασε γρήγορα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έπρεπε πάντα να είμαι ακριβοδίκαιο, αντικειμενικός ε, και αμερόληπτος, να ψάχνω στοιχεία και από τις δύο πλευρές και υπέρ και κατά του προσώπου αυτού. Αυτά λοιπόν ως εισαγγελέα έπρεπε να τα χειριστώ. Και όσον αφορά τα κράτη-μέλη που δεν θα συνεργαστούν με ε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Αυτό ε, θα αφορά φυσικά και το σώμα αλλά και ε, τον Ευρωπαίο εισαγγελέα. Πρέπει να δείξουμε ότι ο Ευρωπαίος εισαγγελέα είναι φορέας, ενδιαφερόμενος και εάν εμφανίζονται προβλήματα θα πρέπει εμείς ως Ευρωπαίοι εισαγγελείς και ο κορυφαίος εισαγγελέα λογοδοτεί απέναντι στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Αυτό λοιπόν θα είναι πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Thank you. And Emilian Pavel for the please. Εμίλιο Πάουλα από το Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που δεν θα έχετε γλωσσικά ζητήματα. Service is regulated differently across... Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι η ρύθμιση είναι διαφορετική. Investigating PIF offenses at national level in equal manner across member states and how do you want to make Πώς θα προωθήσετε λοιπόν την διασυνοριακή διερεύνηση και την ανεξαρτησία σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και αν μου επιτρέπετε μια δεύτερη ερώτηση, ε, Θεωρείτε ότι τα μυστικά πρωτόκολλα με μυστικές υπηρεσίες από διάφορα κράτη-μέλη για την συλλογή μεταφορά πληροφοριών ε, μπορούν να σας βοηθήσουν στις ε, έρευνες σας ή στις έρευνες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σας ευχαριστώ. Εις ό,τι αφορά τη δουλειά του αποσπασμένου εισαγγελέα ή στο γραφείο, θα είναι ένα από τα ισχυρά σημεία της δραστηριότητας ε, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το είπα και το επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω. Θα είναι ο Ευρωπαίος εισαγγελέα η υπηρεσία που θα αναλαμβάνει την σχέση, την επικοινωνία με τα Εθνικά Γραφεία εισαγγελία. Αλλά θα εξαρτάται και από τα κράτη-μέλη να τοποθετούν τον αποσπασμένο του εισαγγελέα σε στρατηγικό σημείο ώστε να μπορεί να διαβιβάζει τις σημαντικές πληροφορίες από τους πιο σημαντικούς φακέλους για, για την εγκληματική δραστηριότητα για την απάτη. Αλλά αν έχουμε δύο ή τρει αποσπασμένου αγγελεί που θα καλύπτουν ένα σημαντικό τμήμα εδάφους, θα πρέπει και αυτοί να είναι σε επαφή με τις ε, ε, εθνικές εισαγγελίε. Επομένω θα χρειαστεί μια τέτοια οργάνωση, μια τέτοια δομή, ώστε να κυλά ομαλά η πληροφορία για να αποφεύγουμε ακριβώς σημαντικά ζητήματα που σήμερα ασκείται κριτική επειδή δεν παρακολουθούνται να εμφανίζονται στην οθόνη του ραντάρ, για να το πούμε έτσι, της ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μια τέτοια δομή θα μας χρειαστεί άμεσα. Τώρα, ρωτάτε γιατί γιατί όλο και περισσότερο βλέπουμε intelligence, δηλαδή πληροφορίες εμπιστευτικές επί συγκεκριμένου πεδίου, να κυκλοφορούν. Εγώ είμαι συνηθισμένο στην Γαλλική Εισαγγελία να ε, συνεργάζομαι με υπηρεσίες που μου φέρνουν αποδείξεις, αποδεικτικά στοιχεία, όχι φήμες και ως Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα πρέπει να κάνω το ίδιο. Η Μόνικα Μακοβέη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτη ερώτηση. Πιστεύετε ότι ο ρόλος του Ευρωπαίου Εισαγγελέα είναι ρόλος συντονιστή, διπλωματικού ε, συντονιστή ανάμεσα στα κράτη-μέλη και όχι τόσο πολύ να ε, ε, ασχολείται με συγκεκριμένες υποθέσεις. Σκέφτομαι ιδιαίτερα υποθέσεις απάτης. Δεύτερη ερώτηση. Τι εγκλήματα εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα πέρα από την απάτη εις βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΦΠΑ. Ε, τι άλλα εγκλήματα εμπίπτουν στη δικαιοδοσία σας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαντήσω επί των δύο αυτών σημείων ως εξής ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αγγελίας θα πρέπει να έχει και τις δύο αυτές ικανότητες. Συντονισμού και διπλωματικής ευαισθησίας βεβαίως, αλλά όχι μόνο. Θα πρέπει να γνωρίζει το πεδίο του. Όταν οι εισαγγελίε θα αναφέρονται σε διασυνοριακή απάντη και ξέπλυμα χρήματος, θα πρέπει να γνωρίζει κανείς το μηχανισμό και τις συνθήκες επί τις οποίες οποιαδήποτε οποιοδήποτε αδίκημα μπορεί να χαρακτηριστεί έγκλημα ή όχι. Χρειάζεται λοιπόν μια τεχνική αριστεία και μάλιστα στο πλαίσιο αυτό υποβάλλω την υποψηφιότητά μου αλλά και βάσει του κανονισμού η PPO από την εισαγγελία θα εξαρτάται να κινητοποιείται αυτός ο μηχανισμός ώστε να συνεργάζεται με όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και με τη συνεργασία των κρατών μελών των συμμετεχόντων και μη. Είναι αυτή η δυτή ε, ειδικότητα που θα πρέπει να έχει η εισαγγελία στην οποία αναφέρομαι από την αρχή. Για τον κατάλογο των ε, αδικημάτων. Όταν μιλούμε για αυτά τα ούτω αποκαλούμε τα δικήματα ΠΕΦ e είναι πάνω απ' όλα απάτε σε ΦΠΑ. Και εκεί ο κατάλογος που δίνεται από τον ΕΠΠΟ απλώς αναφέρεται στην οδηγία η οποία καταλογοποιεί τα δικήματα και εκεί στο πεδίο αυτό έχουμε κάθε είδους αδίκημα. Απάτη, κατάχρηση, κατασπατάληση, ξέπλυμα χρήματος και όλα αυτά θα είναι στο πεδίο ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. E Ο κύριος Ράντεφ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Вие наистина осъзнавате Σας ευχαριστώ λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Έχετε μεγάλη εμπειρία από την Γαλλική Εισαγγελία και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και με την ίδρυση της ε, Eurojust Με συγχωρείτε και πάλι κύριε Ράντεφ. disappoint us, Monsieur Bernard, really, honestly. I mean, really... Имайки предвид вашия богат опит, вие... Λοιπόν, έχετε μεγάλη εμπειρία και γνωρίζετε ποιες είναι οι προκλήσεις ενώπιον της ε, Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Στις απαντήσεις σας μιλάτε για την αναγκαιότητα μιας ισορροπίας, ενός διαλόγου, μιας συνένεσης και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω πώς βλέπετε τον διάλογο και την ε, συνεργασία μεταξύ των εισαγγελιών για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Μιλήσατε επίσης για μια πιθανή δίκευση των διαφόρων ποιμάτων, είτε γεωγραφική είτε κατά τομείς. Και τέλος, τι θα κάνετε έτσι ώστε να γίνει γνωστή η εργασία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στους πολίτες. <laughs> That's only one. Ε, monsieur le député, je, effectivement... Να σας απαντήσω. Σχετικά με την λειτουργία των μονίμων αυτών σωμάτων, ε, πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο και σημαντικό θέμα που θα πρέπει να επιλύσουμε ευθύ εξ αρχή, διότι εντός της δομής της αγγελίας αυτά τα μόνιμα σώματα είναι, θα είναι η κινητήριος δύναμη του τρόπου με τον οποίο θα εξετάζουμε επιχειρησιακά το κάθε Και θα πρέπει ο επικεφαλής να μεριμνεί ώστε η κατανομή μεταξύ των επιμέρους σωμάτων να είναι ίση και βεβαίω θα πρέπει να δούμε και τα θέματα τη σύνθεση των σωμάτων αυτών των εισαγγελικών. Και αυτό θα είναι οπωσδήποτε ευθύνη του επικεφαλή, διότι από εκεί και πέρα όλα αυτά θα έχουν αντίκτυπο επιχειρησιακό μαζί με τον ε, αποσπασμένο εισαγγελέα, το οποίο θα πρέπει από κοινού με το ενδιαφέρομενο κράτο μέλο να διαβιβάσει τι πληροφορίε προ τα άνω και προ τα κάτω τι Εισαγγελικέ ε, διαταγές ε, ε, ερεύνη που θα πρέπει να διαβιβαστούν. Και εκεί η ισορροπία θα είναι πραγματικά πολύτιμη. Ο κανονισμός μας λέει ότι η δουλειά αυτή θα κατανέμεται στην τύχη. Έτσι λέει το, το αρχικό κείμενο. Αυτόν τον παράγοντα τύχης θα πρέπει να τον διορθώνουμε στην πράξη επί τη βάση κριτηρίων είτε λειτουργίας είτε γεωγραφικών. Εγώ θα έλεγα ότι σε πρώτη ε, ανάγνωση θα πρέπει σε τέτοια κριτήρια να βασιστούμε χωρίς να έχουμε προαποφασίσει κάποιους λεπτομέρειες κανόνες. Um, um, Και τελευταία ερώτηση, Τίτμαρ Κώστερ, S&D, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την παρουσίασή σας. Εδώ, εδώ κάθομαι. Συγγνώμη, ναι, βλέπω ότι ε, ε, ο φωτισμός εκεί είναι αρκετά καλός. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπονέρτ, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Η ερώτησή μου έχει ως εξής. Είχατε ποτέ πολύπλοκες διασυνοριακές έρευνες στο πλαίσιο υπερεθνικού φορέα που να απαιτεί συντονισμό διαπραγματεύσεις ε, και επίλυση πιθανών συγκρούσεων δικαιοδοσίας ανάμεσα στις διάφορες εθνικές αρχές ποιο θεωρείτε ότι είναι, ποια θεωρείτε ότι είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να δείξετε την προστιθέμενη αυτή αξία στα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην Εισαγγελία, ώστε να τα ενθαρρύνετε να επιλέξουν συμμετοχή σε μεταγενέστερο στάδιο. Και έχετε εμπειρία από υποθέσεις νομοποίησης παράνομων εσόδων, ξεπλήματος ε, μαύρου χρήματος. Να σας απαντήσω ως εξής σχετικά με τον συντονισμό και την διαπραγμάτευση σε διασυνοριακούς φακέλους. Θα αναφερθώ και πάλι παραδειγματικά στην, ε, ως παράδειγμα μάλλον στην εμπειρία μου από την Eurojust όπου σε φάκελο ακριβώς ξεπλήματος χρήματος και απάτηση δάση, διασυνοριακής, διεθνούς δηλαδή, η οποία αφορούσε σε πέντε χώρες, όχι όλα αλλά μεταξύ των οποίων ήταν και η Ελβετία. Και μέσω της συμφωνίας συνεργασίας που έχει υπογράψει η Eurojust με την Ελβετία, καταφέραμε στο φάκελο εκείνο σε μία μέρα να αποφασίσουμε από κοινού, να συμφωνήσουμε δηλαδή, τις έρευνες σε περί τα δέκα τραπεζικά ιδρύματα μέσα σε μία μέρα και να εκδώσουμε τις σχετικές διαταγές. και στραφήκαμε στον Βέλγο εισαγγελέα ο οποίος ενέχεται και τον ρωτήσαμε πότε θα θέλατε να εκδοθούν οι εντολές αυτές και να διενεργηθούν οι σχετικές έρευνες. Εκείνη την ίδια μέρα ελήφθη η απόφαση, τα μέτρα εφαρμόστηκαν, εκτελέστηκαν και στις πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελβετία, έγιναν οι σχετικές κατασχέσεις και οι σχετικές έρευνες. και το 80% της ε, οικονομικής ζημίας του φακέλου εκείνου που ήταν 10 εκατομμύρια πάγωσε, κατασχέθηκε και επομένως επιστράφει. Εκεί θα πρέπει να αποδείξουμε λοιπόν, να καταδείξουμε αυτήν την ε, προσθέμενη αξία που θα ενέχει το σύστημα αυτό. Και με τέτοια παραδείγματα θα μπορέσουμε να δείξουμε και σε όλους τους υπόλοιπους πόσο σημαντικός θα είναι ο θεσμός. Συνεχίζουμε. Ωραία. Χαίρομαι που σας ακούω, πραγματικά αυτό διαφημίζονται πολύ καλά οι Γάλλοι. Θέλω να σα ρωτήσω για τη σχέση με τον Όλαφ. Ποιον ρόλο βλέπετε για τον Όλαφ και τις διοικητικές έρευνες. Είναι ένα περίεργο θέμα οι διοικητικές έρευνες. Δεν είναι γνωστές σε όλα τα κράτη-μέλη. Έχουμε πάρα πολλά α, προβλήματα. και βεβαίω θα έχετε τη στήριξή μου αν ε, επιθυμείτε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά τις ε, διοικητικές ε, έρευνες, πράγματι είναι ένα ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί θα πρέπει να κάνει δικαστικές έρευνες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το μεγάλο θέμα αφορά ακριβώς τη μελλοντική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Αγγελίας και Όλαφ για να συνεργαστούν οι μεν στην διοικητική πλευρά και η Ευρωπαϊκή Αγγελία στο δικαστικό επίπεδο. Θεωρώ ότι εκεί πέρα πρέπει να υπάρξει κάποια πρόοδος. Είπα ότι είναι μια τεράστια πρόκληση την οποία πρέπει να αναλάβουμε γιατί γνωρίζω βεβαίως ότι στο μέλλον γιατί υπάρχει κάποια σκέψη για μεταρρύθμιση του σχετικού κανονισμού, να ληφθούν κάποιες αποφάσεις έτσι ώστε όλα αυτά να ε, συγκεραστούν κάπως, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπορεί να ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή υπεραξία του Όλαφ και βεβαίως οι διοικητικές έρευνες είναι αναγκαίες ε, όταν έχει νόημα ε, να μιλήσουμε και για την ανάκτηση χρημάτων. Αυτό μπορεί να κάνει ο Όλαφ. Ο Όλαφ έχει επίσης το πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ότι γνωρίζει όλες αυτές τις υποθέσεις, ειδικά το οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν γνωρίζει γιατί δεν υπάρχει. Και υποθέτω ότι στο μέλλον αυτή η διαλειτουργικότητα όπως λέγεται, η δυνατότητα δηλαδή της ε, συνεργασίας θα πρέπει να ενισχυθεί έτσι ώστε η ευρωπαϊκή αυτή εισαγγελία να μπορέσει να προφύσει αυτήν την ε, βαθιά πληροφορία που έχει όλα Όλαφ, να την χρησιμοποιήσει και βέβαια όλα αυτά να μπορέσουν να σταθούν ε, μπροστά σε ένα δικαστήριο. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικότερο. Και ε, να καταλήξουμε σε μια απόφαση. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε μαζί με τον Όλαφ. Σας ευχαριστώ κύριε Σπυρνισκή. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σαφώς ε, κύριε Μπόνερτ ε, έχετε όπως λέτε πολύ μεγάλη πείρα στην ευρωπαϊκή συνεργασία στα ποινικά ζητήματα. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Υπάρχει βεβαίως ε, πράγματι ένας ε, σημαντικός ε, βαθμός διπλωματικής ικανότητας που απαιτείται για αυτά τα οποία κάνετε. Επίσης βεβαίως πρέπει να έχετε και την τεχνική γνώση. Πώς μπορείτε όμως να μας αποδείξετε ότι αυτές οι ικανότητες θα σας κάνουν πιο ε, στιβαρό αν θέλετε και δυναμικό ως εισαγγελέα αντί να προσπαθείτε να βρείτε ε, διευθετήσεις. Ε, δηλαδή πώς θα είστε επίμονος μέχρι το τέλος ε, να φτάνετε των υποθέσεων και να κάνετε κάτι καλύτερο από το να είστε απλά επιθετικός. Κοιτάξτε, ένα εισαγγελέα κατά την άποψή μου δεν πρέπει ποτέ να είναι υπερβολικά επιθετικό. Πρέπει όμω να είναι αποφασισμένο. Και βεβαίω η διπλωματία και τα ωρία τη. Το να είναι κανεί διπλωμάτη σημαίνει να μπορεί να αισθάνεται τα στοιχεία μιας κατάστασης, να αντιλαμβάνεται εφιός την κατάσταση, αλλά μέχρι εκεί. Όταν ο εισαγγελέα είναι στα πλαίσια της αρμοδιότητας και της εντολής του και χρειάζεται να λάβει μια απόφαση, τη λαμβάνει και αυτό έχω κάνει και στο παρελθόν ο ίδιος ως εισαγγελέα της Γαλλικής Δημοκρατίας. Και πάντοτε ήθελα να έχω γύρω μου, ιδιαίτερα για τις δύσκολες αποφάσεις, τους πιο άμεσους συνεργάτες του. Συνεργάτες μου. Και όχι για να κρυφτώ πίσω από αυτούς, γιατί έχω γύρω μου τους πιο αποτελεσματικούς, τους ευφιέστερους ανθρώπους που μπορώ. Βεβαίως, πάντοτε έχω την, το τελικό βάρος της απόφασης. Και δεν θέλω να αφήνω κανέναν από τους συνεργάτες μου να του ρίχνω να μεταβιβάζω το βάρος της απόφασης την ευθύνη πάνω του. Δική μου είναι τελικός. Και πρέπει να είναι και του επικεφαλής εισαγγελέως είναι η ευθύνη. Και ποτέ δεν πρέπει να φοβάται να πάρει την απόφαση που πρέπει να πάρει. Τι λέει ο ποινικό κώδικας, τι λέει η ποινική νομοθεσία στην ε, συγκεκριμένη χώρα, έχει τελεστεί η συγκεκριμένη εγκληματική πράξη. Έχουμε αποδεικτικά στοιχεία. Λαμβάνουμε την απόφαση. Ως 32 χρόνια Ω νεαρός εισαγγελέα και σήμερα ως γενικός εισαγγελέα τα ίδια έκανα. Και ήταν πάντοτε ήμουν αποφασισμένος να μην αποκλίνω ποτέ από τη στόχευσή μου. Η κυρία Μακοβέη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, εξετάζοντας την έκθεση του Όλαφ του 2017, βλέπουμε ότι πολλές ε, έρευνες για απάτη ε, που είχαν να κάνουν με ευρωπαϊκούς πόρους αφορούσαν τη Ρουμανία, 11 συνολικά και μετά είχαμε 12 περίπου Πολωνία-Ουγγαρία και είχαμε την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και σε μικρότερο αριθμό τη Γερμανία, την Ιταλία και άλλες χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Το μέγεθος, οι διαστάσεις της απάτης που έχουν να κάνουν με πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το ΦΠΑ. Ε, το μέγεθος λοιπόν είναι πολύ σημαντικό στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Φαίνεται εκεί να είναι πιο σοβαρό το πρόβλημα από ό,τι σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτό προκύπτει από την έκθεση του Όλαφ. Τι εμπειρίες έχετε λοιπόν όσον αφορά την καταπολέμηση τέτοιων εγκλημάτων, οικονομικών εγκλημάτων, που αφορούν και το πολιτικό επίπεδο. Κάτι που βλέπουμε σε κάποια κράτη-μέλη, που μάλιστα δεν ήταν κράτη-μέλη όταν βρισκόσασταν εσείς στη Eurojust. Μιλάω συγκεκριμένα για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Κοιτάξτε, μεταξύ του 2003 και 2007 όταν ήμουν στη Eurojust ε, είδα, υποδεχθήκαμε τις δύο αυτές χώρες στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε μαζί τους. Υπάρχουν τα μεγέθη στα οποία αναφέρεστε της έκθεσης του 2007 που κατονομάζουν μια σειρά από υποθέσεις με στοιχεία, με μεγέθη, ίσως όχι εξατλητικά. Δεν λέγω ότι τα μεγέθη που έχετε εσείς δεν είναι εξαντλητικά για τις χώρες αυτές, αλλά θα πρέπει να σκεπτόμαστε και τα παλαιότερα κράτη-μέλη, όπως και τη χώρα από την οποία προέρχομαι εγώ. Αλλά ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, οπωσδήποτε δεν θα είναι η εντολή μου να κρίνω κάθε χώρα από τον αριθμό των φακέλων των υποθέσεων που θα την αφορούν. Δεν θα είμαστε εκεί για να καταδεικνύουμε κανέναν ή να ντροπιάζουμε κανέναν. Διότι υπάρχει πάρα πολύ υλικό και πάρα πολλοί φάκελοι που χρήζουν εξέτασης και στην χώρα μου. όπου προέρχομαι από την Βουργουνδία, όπου είναι μια σχετικά ειρηνική περιφέρεια με καλό κρασί, αλλά έχουμε και περιπτώσεις, ειδικά στην ινοκαλλιέργεια, τέτοιες περιπτώσεις που πολλοί από τους συναδέλφους μου στη Γαλλία εξεπλάγησαν με χρηματικές, οικονομικές απάτες λοιπά. Τώρα, μπορεί στην οικονομική απάτη να μην έχω την ίδια εξειδίκευση και την ίδια εμπειρία που έχουν άλλοι υποψηφοί, αυτό το ομολογώ, ωστόσο έχω κάποιες εμπειρίες στο παρελθόν που αυτή τη στιγμή με βοηθούν να αναλάβω αυτά τα καθήκοντα. Η κυρία Ινετφέλτ, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν νομίζω κανείς να αμφιβάλλει αγαπητέ ότι είστε εξαιρετικός εισαγγελέα, όπως είπατε, αλλά το θέμα είναι και το έθεσε και ο συνάλφος των ε, σοσιαλδημοκρατών, εάν ε, ε, πραγματικά μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτή τη δουλειά. Γιατί η απάτη με τα κοινοτικά κονδύλια δεν είναι θέμα να κλέβουμε στον ισολογισμό. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να σκοτώσουν όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Και το πρόβλημα είναι ότι οι κυβερνήσεις δεν είναι απαραίτητα στο πλευρό σας κυβερνήσεις ε, είναι αυτές που θα ερευνήσετε. Είναι τελείως ε, διαφορετικό, διαφορετική υπόθεση. Οπότε το ερώτημα είναι θα βασιστείτε στα στοιχεία που σας δίνουν μόνο τα ή και σε άλλα στοιχεία. Ε, Πράγματι, το θέμα της Αποφασιστικότητα ε, του εισαγγελέα ε, δοκιμάζεται ιδιαίτερα όταν πρέπει να αναλάβει δράση κατά των συγκεκριμένης χώρα μέλου. Αλλά αυτή η εικόνα του ε, Pitbull ίσως ο όρος να φαίνεται λίγο υπερβολικός αλλά χρειάζεται πράγματι μια αποφασιστικότητα και μια ετοιμότητα, δύναμη να αντιμετωπίσει κανείς το έγκλημα ακριβώς και όπως ένα ακριβώς όπως ένα λαγωνικό ή ένα bulldog τέλος πάντων. Και θα πρέπει λοιπόν ο επικεφαλής της Γενικής Εισαγγελίας να αναλαμβάνει δράση όπου θα πρέπει, όπου θα απαιτείται η δράση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και θα πρέπει να αναζητεί και να εξασφαλίζει τη συνεργασία όλων των συμμάχων που θα χρειάζεται. Μεταξύ των οποίων εσείς αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Γενικός Ευρωπαϊκός Εισαγγελίας είναι υπόλογος απέναντί σας. Είναι δηλαδή υπεύθυνο για την δράση και τη δραστηριότητά του απέναντι σε εσά, τα μέλη του Κοινοβουλίου και τελικά τους Ευρωπαίους πολίτες. Και θα πρέπει βεβαίως ο, κάθε εργαζόμενος στην εισαγγελία, ο κάθε εισαγγελέας να αποδεικνύει το θάρρος και την αποφασιστικότητά του. Εγώ σήμερα είμαι μπροστά σας υποψήφιος χωρίς να έχω καμία ανησυχία ή καμία, κανένα φόβο για, το, για την δραστηριότητά μου ως Γάλλου εισαγγελέα στο παρελθόν. Thank you very much. Ευχαριστώ που ήρθατε κύριε Μπονάρτ, εδώ πέρα είμαι. Αναφέρατε στην εισαγωγή σας πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να πείσει τα κράτη-μέλη να ενταχθούν. Καλή τύχη σας εύχομαι. Έχοντας ε, κατά νου ότι ο επικεφαλής εισαγγελίας Ουγγαρίας είπε ότι η Ουγγαρία δεν θα μπει γιατί ε, είναι χαμηλή η ποιότητα. Οπότε είναι δύσκολη η δουλειά σας. Η ερώτησή μου είναι αρκετά ε, πολιτική. Κοιτάξτε. θα ε, ασκείται πολιτική πίεση και σε εσά και εντό των κρατών μελών πώς μπορείτε να προστατεύσετε τους δικούς σας, ε, την ομάδα σας. Και το άλλο ερώτημα είναι αν μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα για την ε, συστημική διαφθορά και κατάχρηση των ε, κοινοτικών κονδυλίων. έχετε δει ποτέ κάτι τέτοιο και τι σκοπεύετε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. Για την πρώτη σας ερώτηση θα έλεγα ότι θα πρέπει ο Ευρωπαίος Αγγελέας να είναι πρότυπο, αλλά δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα πρέπει να ασκεί πολιτική προς τα μη συμμετέχοντα κράτη. Δεν νομίζω ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητά του ή στην εντολή του να πείθει μεμονωμένα το χ ή το ψ κράτος μέλος να εισέλθει στην ενισχυμένη συνεργασία. Δεν τον βλέπω καθόλου έτσι. Νομίζω ότι εκεί υπάρχουν άλλα πεδία, άλλοι υπεύθυνοι για μια τέτοια δραστηριότητα πολιτική. Αλλά και στην Eurojust είχα δει με απόλυτη σαφήνεια συναδέλφους κρατημέλη που ανφίβαλαν και που έλεγαν και τι θα είναι αυτό το πράγμα τι θα κάνει τελικά αυτό το γραφείο η Eurojust δηλαδή. Και δείξαμε με την πράξη μας ότι μπορέσαμε να κερδίσουμε εκείνο το ύψος πορείας που σας έλεγα πριν για το αεροσκάφος και να δείξουμε την προστιθέμενη αξία της υπηρεσίας. Θα χρειαστεί λοιπόν να αποδείξουμε το πόσο πολύτιμη θα είναι η εργασία μας, ώστε να προσελκύσουμε κρατημέλη στην ενισχυμένη συνεργασία. και θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι, Ευρωπαϊ... οι ευρωπαϊκές εισαγγελίες και ιδιαίτερα οι εισαγγελίες οι αποσπασμένοι να προστατεύονται από τις υπερβολικές πιέσεις και εκεί θα πρέπει να εγκαταστηθεί ένας προσωπικός και πολύ στενός διάλογος μεταξύ του επικεφαλής της εισαγγελία, των αποσπασμένων και το σύνολο βεβαίως των εισαγγελέων που θα εργάζονται στην υπηρεσία για να αντιμετωπίζουμε αυτές τις πιέσεις και όταν υπάρχουν τέτοιες πιέσεις θα πρέπει ο επικεφαλής να παρεμβαίνει και ακόμα και να καταγγέλει ένα κράτος μέλος συγκεκριμένο όταν αυτό θα απαιτείται. Κύριε Σωμάτζη. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπονέα, θα έχετε καταλάβει ότι το θέμα της ανεξαρτησίας ε, της εισαγγελία είναι κεντρική σημασία και θυμήσατε την ε, πλούσια εμπειρία σας 32 ετών ή στην Γαλλική Εισαγγελία, χώρα η οποία δεν διακρίνεται για την ανεξαρτησία των σωμάτων εισαγγελία της. Βλέπουμε όμως σήμερα, για παράδειγμα, στον τρόπο με τον οποίο επιβάλλεται ο νόμος στο κίνημα των ε, κίνδυνων γυλαίκων τη δράση που αναλαμβάνει η εισαγγελία. Εσείς λοιπόν με 32 χρόνια εμπειρίας μπορείτε να μας βεβαιώσετε ότι ποτέ δεν υπήρξετε θύμα πολιτικής πίεσης, πίεσης εκ από τα πάνω. Σε 32 χρόνια εμπειρίας λοιπόν σε διάφορες γαλλικές εισαγγελίε σίγουρα θα πέρασαν από μπροστά σας τεράστιες υποθέσεις εμβληματική σημασία. σχετικά με θέματα πολιτικά, διαφθοράς, συσχετισμού οικονομικού και πολιτικού βίου και πώς αντιδράσατε σε αυτές τις περιπτώσεις που έφτασαν στα χέρια σας. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Η ανεξαρτησία του δικαστικού στην Γαλλία έχει εξελιχθεί και της εισαγγελία. Υπήρξαν περιπτώσει στο παρελθόν που εγώ δεν τι είχα ζήσει προσωπικά. Αλλά πράγματι από αυτά που και εγώ κατάφερα να δω υπήρξαν περιπτώσει όπου ασκήθηκε πίεση. Υπήρξαν περιπτώσει όπου το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδινε εντολές ή στα γραφεία της εισαγγελία. Αυτό ριζικά άλλαξε και το υπογραμμίζω από το 2013. Με νέο νόμο που απαγορεύει αυτές τις εντολές. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα το τι συμβαίνει από το 2013 και μετά. Θυμάμαι συγκεκριμένη περίπτωση όπου αναζητούσαμε τις συμβουλές της ε, τεχνικής εγκληματικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατόπιν άμεσον άμεση εντολής, άμεση διαταγής του Υπουργού Δικαιοσύνης. Αυτό ήταν το 14-15 αμέσω μετά τη μεταρρύθμιση του νόμου του 2013 Και τότε η υπηρεσία αυτή αρνήθηκε να μου απαντήσει τότε για να μην θεωρηθεί ότι έδινε εντολή υπό τη νέα νομοθεσία. Εγώ βρήκα την, τις πηγές των στοιχείων που έπρεπε να, τη βρω, να βρω με άλλο τρόπο, αλλά ήθελα απλώς να σας δώσω ένα παράδειγμα του, του τρόπου με τον οποίο επηρέασε τους δημοσίους υπαλλήλου και τους δικαστικούς λειτουργούς μετά την υπόθεση Μουλά, την υπόθεση Μεντβέντιεφ στη Γαλλία, υποθέσεις που δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέρμα τους, διότι έχουμε μπροστά μας ακόμα και θεσμική μεταρρύθμιση που απαιτείται για τις ε, μεγάλες ε, περιπτώσεις ε, διαφθοράς και απάτης. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο στα πλαίσια της ε, γαλλογερμανικής δικαστικής συνεργασίας. Νομίζω ότι είναι και στις απαντήσεις σας ε, στην υπαρθμόν 3, αν δεν κάνω λάθος η απάντηση αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας επιτυχία. Κύριε Μπονέρ, um, um, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρου όλων των Ευρωβουλευτών για την ακρόασή σας εδώ πέρα. Σας ε, ευχαριστώ όλους ε, και για την υπομονή σας ε, και για την πειθαρχία που επιδείξατε κάτι που είναι απαραίτητο σε τόσο μακρές συζητήσεις. Κύριε Πονέρ, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα αξιολογήσουμε την ακρόαση και θα ενημερωθείτε ανάλογα. Σας ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο σας και τη συμμετοχή σας στην ακρόαση αυτή. Το εκτιμούμε. Thank you very much. Dear colleagues, uh, we're... Αγαπητοί συνάδελφοι, κοντεύουμε. Έχουμε τώρα την τρίτη υποψήφια. Ξέρω ότι είναι μια μακρά διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ για την αντοχή σας. Η τρίτη υποψήφια καταφτάνει. Σας παρακαλώ λοιπόν να παραμείνετε εδώ από σεβασμό προς ε, την τρίτη υποψήφια. Θα τη δούμε πολύ σύντομα. Um, Συνάδελφοι, αν θέλετε να κάνετε διάλειμμα, ετοιμαζόμουν να πω, αλλά νομίζω ότι προσέρχεται η υποψήφια. Λίγα λεπτά ακόμα. Υπομονή. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ καθίστε. Σας παρακαλώ να επιδείξουμε τον απαραίτητο σεβασμό απέναντι σε όλους τους υποψηφίους. Παρακαλώ λοιπόν ε, περιορίστε τις μετακινήσεις σας ε, και σας παρακαλώ να σεβαστείτε και τον τύπο. Ε, παρακαλώ μπορείτε να, πάρετε, να βγάλετε μερικές φωτογραφίες αλλά εντός λογικών ορίων. Σας παρακαλώ. Ας ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Διότι θα πάρει τον λόγο η υποψήφια. Παρακαλώ αν μπορείτε να πάτε ε, στην άκρη. Νομίζω ότι βγάλατε αρκετές φωτογραφίες. Όλοι σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ να φύγετε από τη μέση. Σας ευχαριστώ. Okay, colleagues, um... Συνάδελφοι, σας παρακαλώ να περιορίσετε τις μετακινήσεις σας εντός της αιθούση από σεβασμό απέναντι σε όλου του υποψήφιους. Στην αρχή του πρώτου ομιλητή είχαμε αρκετά τέτοια, δεν είναι πολύ δίκιο. Ε, φτάσαμε λοιπόν τώρα στην τρίτη υποψήφια, την κυρία Κοβέση. Θα επαναλάβω την ίδια εισαγωγή που είχαμε και στους άλλους υποψηφίους. Την ε, καλωσορίζουμε εδώ στη συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ και θα σας ενημερώσω ότι Ε, καλούμε τους ε, υποψήφιους ε, να κάνουν μια εισαγωγή 7 λεπτών το πολύ. Θα μετράμε το χρόνο και κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων και απαντήσεων βλέπετε στην οθόνη τον, το χρονόμετρο. Μετά από την εισαγωγή θα μπορέσουμε να έχουμε συνολικά 63 λεπτά ερωτήσεις και απαντήσεις. 14 ερωτήσεις από μέλη της ΛΥΜΠΕ, 7 από την Επιτροπή Ελέγχου του, Προ... του Προϋπολογισμού. Ε... Συνολικά τρία λεπτά για κάθε ερώτηση και απάντηση, δηλαδή η ερώτηση ένα λεπτό και η απάντηση δύο λεπτά. Θα είμαι πολύ αυστηρός όσον αφορά το χρόνο. Υπάρχει διερμηνία, μπορείτε λοιπόν να μιλήσετε στη μητρική σας γλώσσα. Σας παρακαλώ να έχετε κατά νου ότι όλα όσα θα πείτε θα μεταφραστούν, οπότε μην μιλάτε πολύ γρήγορα. Με αυτές τις πληροφορίες θα ήθελα, κυρία Κοβέση, να σας καλέσω να κάνετε την εισαγωγή σας. Σας δίνω το λόγο για το πολύ 7 λεπτά. Good afternoon to everyone. Καλό απόγευμα σε όλους. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την υποψηφιότητά μου. Αρχικά θα μιλήσω αγγλικά Μετά όμως, επειδή είναι πολλοί Ρουμάνοι παρόντες και που παρακολουθούν την ακροασία αυτή, θα μιλήσω ρουμάνικα. Καταρχάς να συστηθώ. Λέγομαι Λόρα Κούβεσι και είμαι εισαγγελέα για πάνω από 23 χρόνια. Το μισό της ζωής μου λοιπόν ήμουν εισαγγελέα. Δουλειά μου είναι να φροντίζω να λειτουργεί δικαιοσύνη όταν παραβιάζεται ε, το ποινικό δίκαιο. Ήμουν Γενική Εισαγγελέα της Ρουμανίας επί 6 χρόνια και ε, εισαγγελέα της, ε, ε, της αρχής κατά της διαφθοράς που είναι γνωστή ως DNA. Είναι, η μόνη, είναι ο μόνος φορέας που έχει την δικαιοδοσία να ερευνά υποθέσεις απάτης με πόλους Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς. Ε, θα είναι μοναδική επαγγελματική ευκαιρία ε, η θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα χαρώ πολύ να συνεχίσω τις εργασίες τόσων ανθρώπων που έκαναν νομικό κείμενο μία ιδέα. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια λειτουργική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πολύ σύντομα λοιπόν θα σας παρουσιάσω το όραμά μου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα πρέπει να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, να ανακτά τα ποσά και να φροντίζει για την εφαρμογή του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα πρέπει να γίνει γι' αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη υποδομή, ε, το ανθρώπινο δυναμικό και ε, η δομή γενικά θα πρέπει να συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη, να ορίζει τους εσωτερικούς κανόνες ε, και τους διοικητικούς κανόνες, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την προστασία δεδομένων, ε, τα ανθρώπινο δυναμικό και τους οικονομικούς κανόνες. Ε, οι εισαγγελεί για να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά θα πρέπει να θέσουν στόχους και στρατηγικές σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εισαγγελεί να καθορίσουμε ε, διαδικασίες για την εφαρμογή των στρατηγικών, ε, ε, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και να συμφωνήσουμε τις προτεραιότητες μας με τις εθνικές αρχές. Θα πρέπει επίσης να έχουμε διευρυμένη συνεργασία με κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν, καθώς και συνεργασία με τρίτες χώρες. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε συμφωνίες σε υπηρεσιακό επίπεδο με την Eurojust, την Europol και με τις ε, κοινέ ομάδες ε, ερευνών ε, και θα πρέπει να εξετάσουμε την τυπολογία τους κινδύνους και τις τροτότητες στις διαδικασίες μας. Πώς μπορώ εγώ να συμβάλλω σε όλα αυτά. Με το καλό παράδειγμα. Έχω εμπειρία στην ε, διαχείριση μεγάλων ομάδων, τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, ε, την ε, έκδοση εσωτερικών κανόνων και κατευθυντήριων γραμμών. Έχω συνηθίσει να δουλεύω υποπίεση και μαζί με την ε, ομάδα μου, μαζί με τους συνεργάτες μου, έχω αυξήσει την αποτελεσματικότητα ερευνών ε, σε περιπτώσεις σοβαρής διαφθοράς. Και η ανάκτηση των πόρων ήταν ε, το επίκεντρο των εργασιών μου. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ έχω ανακτήσει κατά τη διάρκεια του λειτουργήματός μου και ως αποτέλεσμα είχαμε αύξηση των ανακτώμενων ε, ποσών σε 300 εκατομμύρια το, χρόνια, το χρόνο, 10, 10 φορές περισσότερο από ό,τι στα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε δικαστική ε, συνεργασία με πάνω από 40 χώρες, ε, κατάσχεση στοιχείων του ενεργητικού και κατάσχεση λογαριασμών τραπέζι σε άλλες χώρες. μπορώ να λαμβάνω στρατηγικά μέτρα και αυτά είναι τα επαγγελματικά μου επιτεύγματα. Με βάση λοιπόν την εμπειρία μου, ε, ποιες είναι οι αρχές ε, που καθορίζουν τις δράσεις μου. Θα σας τα πω αυτό πολύ σύντομα. Πιστεύω ότι ο εισαγγελέα θα πρέπει να έχει στόχο την αλήθεια. Θα πρέπει να είναι υπηρέτης του κράτους δικαίου και να ε, είναι ηθικά διάβλητος. Θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και απέναντι στο έγκλημα θα πρέπει να εφαρμόζουμε το δίκαιο και να σεβόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα των ε, ανθρώπων που συμμετέχουν στις έρευνες. Και γι' αυτό ε, είναι σημαντική η εισαγγελίση για το κράτος δικαίου. Είναι καθήκον μας να εφαρμόζουμε το νόμο ε, το ίδιο απέναντι σε όλους. Και αυτό ε, αντιπροσώπευαν ε, ο Τζομάν Φραγκόνη και ο Πιέρ Μισελ. Πιστεύω ότι μόνο ένας επαγγελματικό και ανεξάρτητος ε, τομέα δικαιοσύνη μπορεί να καταπολεμήσει το σοβαρό έγκλημα και το οικονομικό έγκλημα. Η ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα δεν είναι προνόμιο για τους εισαγγελείς και του δικαστέ. Μόνο η ανεξάρτητη δικαιοσύνη μπορεί να εφαρμόζει ίσα τον νόμο σε όλους. Επίση, πιστεύω ότι η ανεξαρτησία και η λογοδοσία πάντα πηγαίνουν μαζί. Από την άλλη γνωρίζω ότι έχετε λάβει πολλές αρνητικές πληροφορίες για μένα. Θα ήθελα να πω σαφώς ότι δεν έχω τίποτα απολύτως να κρύψω. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε όλες σας τις ερωτήσεις σήμερα. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, το Κοινοβούλιο έχει αγωνιστεί για να έχει ισχυρό ε, ευρωπαϊκό εισαγγελέα και το Κοινοβούλιο υπερασπίζεται το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Για το λόγο αυτό ε, θα προστατεύσουμε σωστά του οικονομικού πόρου του Ευρωπαίου πολίτη. Σα ευχαριστώ και πάλι που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω την υποψηφιότητά μου και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχω σε μια ανοιχτή και αμερόληπτη διαδικασία κρόασης. Σε ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στις ερωτήσεις. Ξεκινάμε τη Ρομπέρτα Μετσόλα για το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ κύριε Κοβισή που ήρθατε εδώ σήμερα παρά τα δυνατά και πιθανά και απίθανα εμπόδια που έβαλαν στον δρόμο σας. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι και το θάρρος σας πραγματικά απέναντι σε αυτή την επίθεση που έχει εμπνεύσει ανθρώπους όχι μόνο στη Ρουμανία αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ως εισαγγελέα ήσασταν το πρόσωπο τη καταπολέμησης τη διαφθορά στην ε, χώρα σα. Μπορείτε να μα πείτε περισσότερα για την εμπειρία σα για τις ε, γνωστές υποθέσεις σας ε, που βρέθηκαν στο επίκεντρο των ε, ΜΜΕ. Πώς βλέπετε την συνεργασία με τον Όλαφ Όπω ξέρετε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες και πολιτικές ε, υποθέσεις. Έχουμε δει περιπτώσεις ε, ανά την Ευρώπη όπου βλέπουμε τις διοκτικέ αρχές είτε να μην δρούν είτε να μην ερευνούν και να διώκουν ξεκάθαρα ποινικά δικήματα. Τι θα κάνετε με τα κράτη-μέλη που δεν ε, συνεργάζονται. μακροσκελής η ερώτηση, αλλά είναι δύο λεπτά πάντα η απάντηση. Σας ευχαριστώ. Πράγματι, το θέμα των περιπτώσεων που απασχολούν τα μνημεία μπορεί να είμαι σύντομη. Όλες σχεδόν οι περιπτώσεις ε, τις οποίες ερεύνησα είχαν μεγάλο ενδιαφέρον λόγω των ατόμων γιατί η γιατί οι αρμοδιότητες ε, της εισαγγελία μας αφορούν ακριβώς την διαφθορά. Οπότε μιλούσαμε για δημάρχους, ε, επάρχους, ε, γερουσιαστές, βουλευτές, υπουργού, πρώην υπουργούς. Και προφανώς οι πολίτες ήθελαν να μάθουν γιατί ερευνούμε αυτούς τους ανθρώπους. Και πάντα υπήρχε επικοινωνία, σεβόμενη βεβαίως ε, το τεκμήριο της ε, αθωότητας ε, για να προστατεύσουμε τα, τους κατηγορούμενους πάντα σύμφωνα με τους κανόνες που έχει ορίσει το ανώτο το Δικαστικό Συμβουλίο όσον αφορά λοιπόν την εμπειρία που είχα με τον Όλαφ έχω συνεργαστεί και ο κανονισμός επίσης Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι σαφής, μιλάει για στενή συνεργασία με τον Όλαφ και υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχείρισης ε, υποθέσεων. Και υπάρχει και μία διάταξη που λέει πως ε, όταν ξεκινά μία έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Όλαφ δεν θα ξεκινήσει παράλληλα μία έρευνα. Όσον αφορά τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, θα ήθελα να πω πως όπως επίσης προβλέπεται στον κανονισμό θα υπάρχει συνεχής διαβούλευση για ζητήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και επίσης σε σχέση με όλη την δουλειά που γίνεται από τους ε, εντεταλμένους εισαγγελείς και τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Κροβέση, σας ευχαριστώ που ήρθατε, ευχαριστώ και για την τοποθέτησή σας. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε με ποιον τρόπο εξηγείτε πώς ακριβώς θα εκπληρώσετε τα καθήκοντά σας όπως ορίζονται στο άρθρο 14 του κανονισμού ότι δηλαδή θα είστε ανεξάρτητοι πέραν πάσης αμφιβολίας και ότι έχετε τα απαραίτητα προσόντα για διορισμό στα υψηλότερα δικαστικά αξιώματα στο αντίστοιχο κράτος μέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ε, όταν υπέβαλα την ε, υποψηφιότητά μου, βεβαίω ε, διαπίστωσα ότι πληρώ όλα τα κριτήρια όσον αφορά την αρχαιότητά μου σε σχέση με το άρθρο 14 του κανονισμού Ε, το οποίο αναφέρει τα προσόντα, ε, αναφέρει τέσσερις όρους. Πρέπει να υπάρχει αρχαιότητα άνω των 10 ετών, το έχω. Ε, δεν θα πρέπει να έχει υπάρξει συνεργασία με υπηρεσίες πληροφοριών και έχουν γίνει σχετικές δηλώσεις και δεν θα πρέπει να έχει υποστεί ε, πειθαρχικά μέτρα τα τελευταία τρία έτη και να έχει επίσης πολύ καλή αξιολόγηση στην τελευταία αξιολόγησή του. Ε, αυτά τα κριτήρια τα πληρώ μάλιστα ορίστηκα γενικός εισαγγελέας ε, της ε, εισαγγελίας διαφθοράς και έχω και την απαιτούμενη αρχαιότητα για να γίνω εισαγγελέας του ανατάτου δικαστηρίου. Ο νόμος επίσης λέει ότι δεν θα πρέπει να έχει συνεργαστεί κανείς πολιτικά εννοεί με μυστικές υπηρεσίες, όχι την θεσμική υπηρεσία στο πλαίσιο των καθηκόντων του η Χέλγα Στίβενς για το ECR. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα κάνει ε, διασυνεργειακές έρευνες για απάτες ε, για μεγάλα ποσά εις βάρος των ε, κοινοτικών συμφέροντων. Εν τω μεταξύ αυτή τη στιγμή στην ε, Ρουμανία είναι το ζήτημα αυτό ε, πάρα πολύ επίκαιρο. Πώς το βλέπετε και τι ακριβώς θα κάνετε στο ευρωπαϊκό πεδίο. Δεύτερον, υπάρχει μια περίπλοκη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αγγλίας και των κρατών μελών που συμμετέχουν. πώς ε, θα μπορέσετε να αναλάβετε τις υποθέσεις αυτές, τις διασυνοριακές από τα κράτη-μέλη, τα οποία πιθανόν να μην θέλουν ε, είτε να συνεργαστούν είτε και να ασκήσουν πίεση προς την ε, αντίθετη κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε όλες μου τις δραστηριότητες ως γενικός εισαγγελέας, γενικός εισαγγελέας με συγχωρείτε, ως εισαγγελέας μάλλον, στην Ρουμανική εισαγγελία, σεβόμουν όλες τις διατάξεις νομοθεσίας, έπρεπε να είμαι αντικειμενική όπως κάθε άλλος εισαγγελέα και ήμουν αποφασισμένη και θαραλέα. Θεωρώ ότι αν μου δοθεί η ευκαιρία αυτή, όπως έχω πράξει και στο παρελθόν, θα δρώ απολύτως επαγγελματικά σεβόμενοι τις υποχρεώσεις ε, που ε, ε, εξηγούν οι διατάξεις του κανονισμού EPPO και, τον, και οι υπόλοιπε νομοθετικές διατάξεις. Για μένα δεν είναι σημαντικό τι ακριβώς συμβαίνει στη Ρουμανία αυτή τη στιγμή και ποιες ανταλλαγές υπάρχουν μεταξύ Δικαστικού Σώματος και Υπουργείου Δικαιοσύνη. Εγώ πάντοτε θα σεβόμουν τις διατάξεις του κανονισμού εφόσον, ήταν εφόσον θα μου επιτρέπατε να διοριστώ σε αυτήν την ε, θέση. Η Σόφη Ιντεφέλτ για το Άλντι. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε κυρία Τσεβεσί. και μάλλον. Θα ήθελα να εμείνω λίγο περισσότερο στην ερώτηση της κυρίας ε, Στίβενς. Πώς θα χρησιμοποιούσατε συγκεκριμένα νέα, το νέο δίκτυο συντονισμού της Eurojust, ώστε να εξασφαλίσετε ότι τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη όχι μόνο δεν θα παρεμποδίζουν τη δουλειά της αγγελίας, αλλά θα προσεγγελικέται και νέα μέλη. Και δεδομένου του συγκεκριμένου βιογραφικού σας, πώς θα εξασφαλίζετε ότι με αυτή τη συγκεκριμένη δομή που θα έχει και τους αποσπασμένους που θα έχει εισαγγελείς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα γίνει πραγματικά ανεξάρτητο ευρωπαϊκό όργανο και όχι και δεν θα υπάρχει τις κράτη-μέλη και την πίεσή τους. Είναι αλήθεια ότι οι εντεταλμένοι εθνικοί εισαγγελείς θα συνεχίσουν να είναι εισαγγελείς στο πλαίσιο του εθνικού του συστήματος που έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τις αρχές. Ωστόσο, έχουν γίνει διασυνοριακές έρευνες ε, στο παρελθόν και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ολοκλήρωσής τους ήταν η κοινέ ε, ερευνητικέ ομάδε μέσω τη Eurojust, που είναι πολύ αποτελεσματικό μέσω συνεργασία. Αυτό το είδαμε στο παρελθόν αλλά και με την εφαρμογή του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναμένεται από την Eurojust να ε, συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό καθορίζεται σαφώς στην, ε, στον κανονισμό. Επίσης ε, θα υπάρχει υποστήριξη όσον αφορά την παροχή πληροφοριών. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα να Χρησιμοποιούνται τα σημεία επαφής, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσον αφορά τα κράτη-μέλη αυτά που δεν συμμετέχουν, νομίζω ότι εναπόκειται στον Γενικό Εισαγγελέα να ε, συνάψει συμφωνίες με τις εισαγγελίες αυτές και να δημιουργήσει σημεία επαφής κέντρα επαφής. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν μπορούν ε, να λάβουν κίνητρα για υπογραφή των συμφωνιών, αυτών ή ακόμη και ε, να προσχωρήσουν στην εισαγγελία εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει σωστά και ότι είναι αποτελεσματικός φορέας και ότι προστατεύει ε, τα οικονομικά συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Η Εύα Ζολή από τους Πρασίνου, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στην Λάουρα Κοβέση και σε όλους σας ότι είμαι πολύ περήφανη που βρίσκεται εδώ σήμερα, παρά την εκστρατεία που έχει ξεκινήσει εις βάρος της η κυβέρνησή της. Και θα ήθελα να σας πω ότι δεν πιστεύουμε αυτά που υπόθηκαν. Και εγώ προσωπικά έχω ιδιαίτερους λόγους να μην τα πιστεύω όλα αυτά, διότι γνωρίζω πολύ καλά τι συμβαίνει όταν διανεργεί κανείς έρευνες ε, εις βάρος σημαντικών προσώπων ή των δομών της εξουσίας. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην λάβετε υπόψη σε αυτή την εκστρατεία. Και θα ήθελα τώρα να ρωτήσω την Λάουρα Κοβέση τι μέτρα θα αναλάβετε για να διασφαλίσετε τα θεμελιώδη δικαιώματα κατηγορουμένων στο μέλλον, εάν ε, λάβετε τελικά τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα. Μία από τις βασικές ε, αρχές ε, στις οποίες στηρίζεται η Γενική Εισαγγελία είναι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που συμμετέχουν στις έρευνες. Αδιαμφισβήτητα λοιπόν αυτό θα αποτελέσει προτεραιότητα για όλους όσους συμμετέχουν στις εργασίες της εισαγγελία. Επίσης μπορώ να σας πω ότι ως γενική εισαγγελέα στο DNA σε πολλές περιπτώσεις είδα εισαγγελείς που ε, εργάζονταν ε, κατά τη διάρκεια της ε, δικής μου θητείας δέχτηκαν επιπλήξεις σε περίπτωση μη σεβασμού των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. Εάν ως Γενική Εισαγγελέα διαπιστώσω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παραβιάσει τα δικαιώματα κατηγορουμένων, θα φροντίσω να αναλάβω μέτρα για να αποφύγουμε τέτοιες ε, καταστάσεις στο μέλλον. Πολύ σημαντικό όμως είναι εδώ να υποθεί ότι στη Ρουμανία οι εισαγγελείς ελέγχονται από τους δικαστές και ο τρόπος που εργάζονται, ο τρόπος που χειρίζονται αποδεικτικά στοιχεία εποπτεύεται από τους δικαστές. Ως Γενική Αγγελέας και Επικεφαλής του DNA πάντα ήλεγχα τι γίνεται και ρωτούσα τους δικαστές σε περίπτωση που ένας δικαστής ε, θεωρούσε παράνομα ε, μη αποδεκτά τα αποδεκτικά στοιχεία. Ε, φροντίζαμε να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, είμαι εδώ, κυρία ο εφέση ήθελα να εκφράσω την απόλυτη συμπαράστασή μου απέναντι στις επιθέσεις που υφίσταστε και συγκινούμε που αναφέρεται το όνομα του Τζοβάνι Φαλκόνε με τον οποίο εγώ είχα συνεργαστεί προσωπικά στο παρελθόν. Τώρα θα ήθελα μια διευθύνηση από σας. Ε, στις απαντήσεις σας λέτε, αναφέρεστε μάλλον σε δύο τιμητικές, ε, τιμητικούς τίτλους που έχετε λάβει από πλευράς της CIA το 2011 και το 2007 αναγνώριση εξαιρετικής ε, συνεργασίας και υποστήριξης προς τις ε, μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ ήθελα να μου το διευκρινίσετε αυτό. Περί τίνος πρόκειται όταν γράφει κανείς κάτι τέτοιο στο βιογραφικό του σημείωμα. Εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω. Επαναλαμβάνω, είναι 2007 και 2011. Και από το 3 ως το 5 θυμίζω ότι στη Ρουμανία υπήρχαν φυλακές της CIA. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Να κάνω μία διόρθωση. Αυτή δεν ήταν τιμητική, τιμητικές διακρίσεις από την CIA, αλλά από έναν οργανισμό επιβολής του νόμου μυστικές υπηρεσίες στην πραγματικότητα, με διτή αρμοδιότητα να προστατεύει την ασφάλεια των ε, Αμερικανών υπηκόων αλλά και την ε, δημοσιονομική και νομισματική ασφάλεια. Εγώ ως επικεφαλής της Ρουμανικής ε, Εισαγγελίας κατά της διαφθοράς της DNA ε, είχα ερευνήσει μία σειρά από περιπτώσεις για πλαστογράφηση δολαρίων αλλά και για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Ήμουν λοιπόν ένας από τους πρώτους εισαγγελικού στην Ρουμανία που ερευνήσαμε περιπτώσεις phishing γιατί στη Ρουμανία έχουμε ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα ε, με εγκλήματα του ίντερνετ και του κυβερνοχώρου. Τώρα για την προσωπική μου συμμετοχή ε, σε κάποια προγράμματα κατάρτισης ε, και στην υποστήριξη, ενδυνάμωση των εισαγγελικών υπαλλήλων ε, ερευνούν αυτές τις ε, περιπτώσεις ε, απάτης εγκλημάτων στο ίντερνετ. Μου έδωσαν αυτές τις μερικές διακρίσεις οι Αμερικανοί. Ως Γενική εισαγγελέα από το 2 το 7 ασχολήθηκε η εισαγγελία για πρώτη φορά με αυτά τα κρούσματα στην στο ίντερνετ και χρειάστηκε να καταρτιστούν νέοι εισαγγελεί. και για αυτήν τη δουλειά που έκανα στην κατάρτιση νέων εισαγγελέων μου έδωσαν ε, μια διάκριση. Δεν ε, μου προσέφεραν την αμερικανική υπηκότητα, ούτε είμαι βέβαια υπάλληλος της CIA όπως κυκλοφορεί ως φήμη, όλα αυτά είναι ψέματα. Ο κύριος Ιβαν για τους ανεξάρτητους ευχαριστώ πρόεδρε Κυρία Κιόβεση, σε αυτές τις ε, δύο επιτροπές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, μιλούμε για πολύ σημαντικές αξίες για την ανεξαρτησία της εγκαλαικής αρχής, για μηδενική ανοχή στη διαφθορά, το δικαίωμα της έκφρασης, της γνώμης, την ελευθερία του τύπου, την ηθική ακεραιότητα κτλ. κτλ. και το Συμβούλιο εξέδωσε κάποιες συστάσεις ε, σύμφωνα με τις οποίες οι μυστικές υπηρεσίες δεν θα πρέπει να ενέχονται στις ε, ε, υποθέσεις του δικαστηρίου, στις δικαστικές υποθέσεις. Θα είχα λοιπόν στο πλαίσιο αυτό τις εξής ερωτήσεις προς εσάς. Ε, ε, είναι αλήθεια ότι το Δικαστικό Συμβούλιο ε, της Ρουμανίας ε, σημείωσε ότι η εισαγγελία DNA της οποίας Γίστο επηρέασε, παρενέβη μια υπόθεση που ήταν της προσωπικής σας αρμοδιότητας. Δεύτερον, οι ρουμανικές μυστικές υπηρεσίες ήταν πράγματι μέρος κοινών ερευνητικών ομάδων σχετικά με αποδεικτικά στοιχεία των φακέλων που ερευνούσατε. Επίσης, Πώς εξηγείτε ότι το 4% των εισαγγελικών υπαλλήλων που κατηγορήθηκαν κατέληξαν σε απαλλαγές. Κοιτάξτε, εντό δύο λεπτών που είναι πολύ λίγο χρόνο, θα κοιτάξω να σας, θα προσπαθήσω να σα δώσω μια πλήρη απάντηση. Η πράγματι υπήρχε, υπήρξε ε, η εξέταση διαφόρων ε, ψευδών καταγγελιών που έγιναν ε, ε, σε ένα χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών αποδείχθηκε ότι τελικώς ε, τα στοιχεία που είχαν δοθεί ήταν ψευδή. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η περίπτωση διήρκεσε, η έρευνα αυτή διήρκεσε τέσσερα χρόνια. Ε, πολλοί δικαστικοί υπάλληλοι ενέχοντος στην περίπτωση αυτή και σε καμία περίπτωση δεν ενεπλάκην εγώ σε κανενός είδους προσπάθεια επιρροής. Πάρα πολλές ε, δικαστικές αρχές σε διαφορετικά επίπεδα στη χώρα ε, εξέδωσαν πορίσματα υπέρ μου. Εάν το ανώτο δικαστικό αυτό συμβούλιο θεωρεί ότι υπάρχει, ε, ότι ασκήθηκε επιρροή, και παρότι οι δικαστικοί που ενέχονται στις υποθέσεις ε, ε, έχουν δηλώσει ενόρκως ότι σε καμία περίπτωση δεν επηρεάστηκαν από μένα και εκρε, εκρεμούσεις της από το ανώτατο συνταγματικό και ακυρωτικό δικαστήριο στη Ρουμανία και καθότι ενέχονται και άλλα και άλλοι συνάδελφοι και άλλα μέλη της αγγελίας της, κατά τη διαφθοράς ε, είναι λίγο παραπλανητικό να θέτει κανείς το ζήτημα με τον τρόπο που το θέτεται. Επίσης, για τη δεύτερη σας ερώτηση, έγιναν κάποιες ε, παραπομπές ε, ε, που συμπεριελάμβαναν στοιχεία που είχαν ληφθεί από τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά οποιοδήποτε σώμα επιβολής του νόμου υπό την Ρουμανική ε, νομοθεσία υποχρεούται να παράσχει στοιχεία στη δικαιοσύνη. Τα στοιχεία λοιπόν ζητήθηκαν από την εισαγγελία και εξακριβώθηκαν από αυτήν. Κοιτάξτε, ήσασταν πολύ σύντομοι, δεν βλέπω να υπάρχει κανένα πρόβλημα αν έχετε να πείτε κάτι έτσι σύντομα. Ε, σας ευχαριστώ. για το ποσοστό αθώσης 40% ε, δεν ισχύει αυτό. Αυτό δημοσιεύεται κάθε χρόνο. Ήταν μεταξύ 10 και 13%. Μάλλον αναφέρεστε στην τελευταία έκθεση δραστηριοτήτων που δημοσιεύτηκε αυτήν την εβδομάδα. Εκεί πέρα υπήρχε ένα ποσοστό αθώσης 36%. Αλλά εγώ εδώ και 6 μήνες δεν είμαι ε, μέλος αυτής της αγγελίας. Διάβασα την ε, έκθεση αυτή. Μιλάμε για ένα 13,6% πραγματικό ποσοστό αθώσεων. Ε, τεράστια διαφορά από το 36% γιατί πρέπει να δείτε και τις αθωώσεις που αφορούν ε, κάποιες περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας. Λοιπόν, 13% αθώσεων ήταν για άλλες περιπτώσεις και πάνω από 20% των ατόμων που αθωώθηκαν ε, είναι εντός του 3% που έγινε λόγω αποποινικοποίηση ε, των ε, επίμαχων πράξεων. Σα ευχαριστώ. Λοιπόν, για το ΕΛΚ τώρα. Έγγελ, Αγκουάρνου και Ράντεφ. Ποιο είναι? ποιο θα ρωτήσει τελικά. Ο κύριο Αγκουάρνου, παρακαλώ. Τρία ονόματα μου έχουν σημειώσει εδώ, γι' αυτό. Όχι, εγώ ένα όνομα έχω όμω. λέει ο κύριος Ουγγουρεάνου. Ο κύριος Ουγγουρεάνου. Καλησπέρα σας ε, κυρία Καδέση. Ε, οφείλω να σε ρωτήσω ε, το εξή. Το έχουμε ακούσει βεβαίω πολλές φορές, αλλά πρέπει να επιμείνω. Ίσως υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς και η Ρουμανία θα προτείνει τουλάχιστον δύο άτομα για αυτήν την θέση. Αν το αναφέρατε αυτό στις γραπτές απαντήσεις σας. Ε, ίσως υπάρξουν προβλήματα αρχής ε, σε σχέση ακριβώς ε, με το ότι υπάρχουν σε δύο υπηρεσίες και ίσως υπάρχουν αντιφατικές οδηγίες. Το δεύτερο θέμα είναι ότι υπάρχει μια εξαιρετική αλλά υπαρκτή κατάσταση στην Ρουμανία, όπου η κυβέρνηση η οποία θα προτείνει ε, τους ε, εντεταλμένους ε, είναι ανοιχτά εχθρική. Οπότε το ε, ερώτημά μου το εξή πώς θα το επιλύσετε αυτό όσον αφορά τη δουλειά που κάνετε και την εικόνα που μεταδίδεται προς τα έξω. Θα χρησιμοποιήσετε κάποιες εσωτερικές διαδικασίες που θα καταρτήσετε η ίδια ή θα υπάρξει άλλο ένα επίπεδο διαδικασιών. Πώς θα το επιλύσετε αυτό ή τουλάχιστον πώς θα προσπαθήσετε να περιορίσετε τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση και σας ευχαριστώ που επαναλαμβάνετε αυτή την ερώτηση και έχω την ευκαιρία να απαντήσω. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι σύντομος. Όταν μιλάμε για τις δραστηριότητες των εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οδηγίες πάντα δίνονται από τα μόνιμα τμήματα του δικαστηρίου. Και βεβαίως υπάρχει και ο επικεφαλής εισαγγελία και γίνεται μια τυχαία διανομή. Όταν μιλάμε λοιπόν για τους εντεταλμένους ευρωπαϊκούς εισαγγελίες που θα βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη, δηλαδή το ότι ε, συμβαίνει στα μόνιμα τμήματα. Επίσης θα υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Αγγελίας και Εθνικών Αρχών και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στον κανονισμό. Γεγονός είναι πως η κυβέρνηση είναι εχθρική, ειδικά στο πρόσωπό μου. Αλλά δεν θα έπρεπε να είναι εχθρική σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο πρέπει να υπάρχουν τρει εισαγγελίε από την ε, Ρουμανία. Οι κανόνες είναι σαφεί όσον αφορά τι αρχέ των κρατών μελών ε, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα υπάρχει και ένα εσωτερικό κανονισμό που θα εγκριθεί. Φαντάζομαι τώρα δεν μπορώ να σα δώσω κάποιε λεπτομέρειε γιατί ε, αυτό θα εγκριθεί από το Συμβούλιο Ευρωπαίων Εισαγγελίων με πλειοψηφία δύο τρίτων. Οπότε πρώτα πρέπει να συζητηθεί και να διαμορφωθεί από τι συζητήσει με του άλλου Ευρωπαίου Εισαγγελεί και τις εθνικές αρχές, αλλά οπωσδήποτε οι πτυχές αυτές θα πρέπει να εξεταστούν εν καιρό. Ανεξαρτήτως λοιπόν το εάν είναι φιλική ή εχθρική η κυβέρνηση, ο εισαγγελέα πρέπει κανείς να κάνει τη δουλειά της και να σέβεται τα όσα ορίζει ο νόμος. Σας ευχαριστώ κυρία Γκραπίνη για τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Η σχέση ανάμεσα ε, στους ε, διάφορους φορείς διαφέρει στα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, πώς λοιπόν θα εξετάσετε το ρόλο των εντεταλμένων εθνικών εισαγγελέων στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν ήσασταν πολύ ακριβείς όταν αναφερθήκατε σε αυτό πριν. Ε, το CSM σας έχει απαντήσει όσον αφορά την ε, προηγούμενη ε, εμπειρία σας. Πώς μπορείτε όμως να παρακάμψετε αυτό το πρόβλημα της κατάχρησης της θέσης σας, διότι σας απέλησαν από το DNA. Πώς το εξηγείτε αυτό. Μέχρι τώρα δεν είχαμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Σας παρακαλώ να συνεχίσουμε έτσι. Παρακαλώ, μπορείτε να απαντήσετε. Δεν θα έχουμε άλλες τέτοιες παρεμβάσεις, διότι σεβαστήκαμε και τους προηγούμενους υποψηφίους. Σας παρακαλώ λοιπόν να σεβαστείτε και τούτη την υποψήφια. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ ο ενεργός ρόλος ε, του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και των εντεταλμένων εισαγγελέων ε, ε, θα λειτουργήσει σύμφωνα με το Συμβούλιο Ευρωπαίων Εισαγγελέων και τους εσωτερικούς κανόνες που θα θεσπίσει το Συμβούλιο. Όσον αφορά την προηγούμενη πείρα, δεν γνωρίζω τι έχει πει το CSM, αλλά υπάρχει διάταξη που δεν έχει καμία σχέση με την ε, προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία. και άλλοι γενικοί ε, εισαγγελείς και άλλοι στην αρχή μου ε, έλαβαν ε, σχετική απάντηση από το CSM. Υπήρχαν άλλες 7 ε, ε, περιπτώσεις όπου αναγνωρίστηκε η εμπειρία. Μόνο στη δική μου περίπτωση δεν έγινε αυτή η αναγνώριση. Ορίστηκα επικεφαλής του DNA χωρίς να έχω αναγνωρισμένη προηγούμενη εμπειρία. Όσον αφορά την ανάκληση των αρμοδιοτήτων μου, αυτό ήταν αποτέλεσμα Απόφαση ε, του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ε, εγώ δεν είχα καμία σχέση με αυτή την απόφαση. Ε, το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση. Εγώ δεν συμμετείχα στη διαδικασία αυτή, δεν είχα τη δυνατότητα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, ούτε να ασκήσω έφεση για το λόγο αυτό. Έστειλε ένσταση στο Ευρωπαϊκό προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία εξετάζεται αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Αλλά η προσφυγή μου είναι θέμα αρχής. Εάν η εισαγγελεί στη Ρουμανία πρέπει να είναι ε, ε, ε, δεν θα πρέπει απλά να μπορεί να ε, απολυθεί ένας εισαγγελέας από το Σταγματικό Δικαστήριο. Κύριε Μακοβέη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λυπούμε που η πλειοψηφία των ερωτήσεων που απευθύνεται στην υποψήφιο δεν αφορά την εμπειρία της και την εξειδίκευσή της, αλλά τις ε, φήμες απάτης και τις ψευδείς κατηγορίες που κυκλοφορούν κατά του προσώπου σας. Εν εγώ έχω κάποιες πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις για σας. Πώς θα χρησιμοποιήσετε την εμπειρία σας για την καταπολέμηση της διαφοράς. Μήπως ε, θα σας βοηθήσει σε αυτό η ηγεσία της DNA στη Ρουμανία και πώς αντιμετωπίσατε στην εμπειρία τη ρουμανική σας στις ε, τις πολιτικές πιέσεις που σας ασκήθηκαν, γιατί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιστέψτε με, ασκούνται πιέσεις. Τώρα, έχουμε περιπτώσεις απάτης εκατοντάδων χιλιάδων, ε, ε, μάλλον πολύ, υψηλών, πολύ σημαντικών ποσών ε, στην Ανατολική Ευρώπη και μιλούμε για συστημική διαφθορά και συνεχείς συστηματικές παρεμβάσεις των Υπουργείων Δικαιοσύνης σε ιδιαίτερα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στη Ρουμανία. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα της δικής σας δραστηριότητας για την καταπολέμηση των φαινομένων αυτών. Πολύ σύντομα λέει η κυρία Κιόβεση. Ε, κοιτάξτε, για τους ε, φακέλους ε, που εξετάζονται για το όνομά μου είμαι αθώα. Τώρα, για την... για τις περιπτώσεις που αφορούν και σε τρίτες χώρες μπορώ να σας δώσω πρόσθετα στοιχεία εφόσον απελευθερωθούν τα στοιχεία αυτά και εφόσον τα επιθυμείτε. Τώρα μπορώ να σας πω ότι κάθε χρόνο η DNA καταδίκαζε περί τους χίλιους εγκληματίες. Εν πάση περιπτώσει κατά μέσον όρων 900 νομίζω κάθε χρόνο ε, για κάθε χρόνο που ήμουν επικεφαλής της ΔΕΝΑ στη Ρουμανία. Μεταξύ των οποίων είχαμε πρώην υπουργού, γερουσιαστέ, υφυπουργού κτλ. Για τις ε, πολιτικέ πιέσει ε, ως επικεφαλής της εισαγγελία κατά τη διαφορά αλλά και γενική γενικής εισαγγελέα στη Ρουμανία, κάθε φορά που μας καλούσε ένας πολιτικός ή εμένα καλούσε ε, ε, για να ασκήσει πιέσεις, όλα αυτά τα δημοσίευα απευθεία. Τις πληροφορίε αυτές τις έδινα στον τύπο. Και γι' αυτό έπαψαν να προσπαθούν να με καλέσουν. Υπήρξαν άνθρωποι που είχαν σημαντικούς θόκου στην Ρουμανική κυβέρνηση, υπήρξαν εξωτερικέ πιέσει, αλλά κάθε φορά ε, εγώ αντιμετώπιζα το θέμα αυτό και έχω σημαντική εμπειρία ε, Αντιμετώπιση αυτή τη πολιτική πίεση για τι περιπτώσει διαφορά κατά των ευρωπαϊκών πόρων. Κάθε χρόνο που ήμουν ε, στην, ε, στην εντολή αυτή και από την έκθεση του Όλαφ του 2007 και μετά γνωρίζω ότι περί τις 200 περιπτώσεις άνοιγε και έκλεινε κάθε χρόνο η Όλαφ. Κάθε χρόνο. Ίσως αυτό να μην είναι επαρκή σύγκριση, αλλά ήθελα απλώ να σας δείξω ότι απέναντι σε ένα τόσο σημαντικό αριθμό φακελών γνωρίζουμε την μεθοδολογία ε, των εγκληματικών αυτών πρέξενων γνωρίζουμε τις ε, ροές ε, τα ψευδή ή πλαστά έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να υποστηρίξουν αυτή την απάτη και την κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων. Γνωρίζουμε την τυπολογία των περιπτώσεων αυτών, γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο διαπράττονται αυτέ οι πράξεις. Διακόπτει ο πρόεδρο γιατί, ε, με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να ακούσουμε όλα τα μέλη και όλους τους υποψηφίους. Ε, πρέπει να είμαστε πιο ε, πειθαρχημένοι. Ε, ο κύριος Άντρης Μάμεκίνης για τους SND. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητή υποψήφια. Στην, στο πλαίσιο περίπλοκων διασυνοριακών ερευνών Ιδιαίτερα ένα υπερεθνικό σώμα που θα χρειαστεί συντονισμό, διαπραγμάτευση, επίλυση ε, αποκλήσεων ε, μεταξύ των νομοθετικών διατάξεων των χωρών που θα ενέχονται. Τι θεωρείτε ότι θα είναι η προσθέμενη αξία του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία και πώς ε, προτίθεστε να αποδείξετε την ε, προσθέμενη αυτή αξία στα χώρα, στις χώρες εκείνες που δεν έχουν προσχωρήσει στον θεσμό της εισαγγελία ώστε να τις προσελκύσουμε σε μελλοντικό χρονικό σημείο. Σα ευχαριστώ. Ε, στην ε, εισαγγελία κατά της διαφθοράς στη Ρουμανία πράγματι είχαμε πάρα πολλές διασυνοριακές περιπτώσεις και κοινέ επιχειρήσεις ε, με άλλες χώρες όπου ζητούσαν δικαστική αρρωγή μέχρι την περίοδο του 2017 είχαμε περί τις 18 διασυνοριακές τέτοιες περιπτώσεις όπου μας ζήτησε ε, συνεργασία και βοήθεια άλλο κράτος μέλος και είχαμε προχωρήσει σε κατασχέσεις ε, και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και σε άλλες χώρες. Είχαμε διαφορές ε, αποκλήσεις τέλο πάντων ε, ε, νομοθετικών διατάξεων τις οποίες επιλύσαμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και στην κανονισμό EPPO υπάρχει διάταξη σύμφωνα με την οποία κάθε στοιχείο που αφορά σε, άλλη, ε, σε αρμοδιότητα και νομοθεσία άλλης χώρας θα πρέπει να επιλύεται υπό την νομοθεσία της χώρας εκείνης. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια προσέγγιση ώστε να ερευνούμε περιπτώσεις ε, διασυνοριακής απάτης και εγκληματικής δραστηριότητας. Και θα έχουμε και μια ε, εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων στην χώρα που θα ενέχεται και υπό τη δική της νομοθεσία και σε σχέση με διασυνοριακές ε, περιπτώσεις και με αταχύτατη ανταλλαγή πληροφοριών. Άλλο ένα πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι βλέποντας τα διάφορα είδη περιπτώσεων και εγκληματικών πράξεων θα μπορούμε γρήγορα να εντοπίζουμε ε, ελλείμματα ε, και κινδύνους στη διαδικασία ιδιαίτερα για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών πόρων. Και η απάτη με τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν είναι κάτι που θα πρέπει μόνο να ερευνούμε αλλά και να αποτρέπουμε και αυτή η ανάλυση από αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον που εγώ είχα δει θα ήταν εξαιρετικά υψηλής χρησιμότητος. Ευχαριστώ. Ναι, θα μιλήσω γερμανικά. Είμαστε από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Σας ε, γνωρίζουμε, σας εμπιστευτήκαμε στην Ρουμανία και στο ρουμανικό σύστημα για να διώξετε περιπτώσεις ε, ποινικέ και απάτης ε, Βλέπουμε πως όλοι οι υποψήφοι είναι πολύ ικανοί, αλλά εσείς επιπλέον δεν είστε μόνο οι νεότεροι, αλλά και ικανότατοι, οπότε λυπούμε πράγματι για αυτά τα οποία ακούστηκαν, γιατί ε, σας χρειαζόμαστε τελικά σε αυτήν την σημαντική θέση. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα που αφορά τις ε, διοικητικές έρευνες ε, του Όλαφ. Ποια σχέση βλέπετε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ είμαι εισηγήτρια για τον κανονισμό του Όλαφ. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Όπως είπα, έχω συνεργαστεί στενά με τον Όλαφ και ο ρόλος των διοικητικών ερευνών ήταν ακριβώς ένα πρώτο βήμα στην ποινική έρευνα. Όλες αυτές οι διοικητικέ εκθέσεις όμως, τουλάχιστον στις έρευνες στις οποίες είχα εμπλακεί εγώ, είχαν ολοκληρωθεί με διοικητικά στοιχεία που μετά εντάχθηκαν στην ποινική διαδικασία και για τους ε, κατηγορούμενους και για τους ε, υπόλοιπους. Όσον αφορά λοιπόν τη συνεργασία με τον Όλαφ, θεωρώ ότι θα πρέπει να περιορίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών. Και οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ε, δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνονται με διοικητικέ έρευνε ε, του Όλαφ. Η προτεραιότητα, και αυτό παρουσιάζεται στον οργανισμό, θα πρέπει να είναι να δράσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν συμβεί αυτό, μπορεί να υπάρξει παράλληλα και διοικητική έρευνα του Όλαφ, ο οποίο όμω μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση τη απάτη με ευρωπαϊκά κονδύλια και στην ε, δουλειά που κάνει σε σχέση με την καταπολέμηση της ε, απάτης. Ειδικά για περιπτώσεις οι οποίες ε, δεν αφορούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σας ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ. Ναι, σας ευχαριστώ. Η κυρία Κιόβεση και εγώ λυπούμαι για τις πιέσεις που σας ασκούνται. Δεν θα αναφερθώ τώρα για πιάσεις που ασκούνται στις, ε, στους ε, Ισπανούς εισαγγελείς και δικαστικούς, ε, γιατί εξορισμού έχουμε αυτά τα προβλήματα. Από την άλλη μεριά επίσης εξορισμού η εισαγγελία πρέπει να είναι εξάρτητη. Τώρα, έμπασε ρητώσει Εσείς ε, νομίζω ότι το 2017 ε, λάβατε ένα παράσημο από την ε, Χάνσα που είναι ένα, ε, ένας θεμελιακός θεσμός και νομίζω ότι ήδη λάβατε μάλλον για όλε τι κατηγορίε που ακούγονται οπωσδήποτε δεν διευκόλυναν το έργο σα ούτε την υποψηφιότητά σα τη σημερινή. Τώρα πώς μπορείτε, αυτή είναι η ερώτησή μου, πώς μπορείτε να συνεργαστείτε με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εισαγγελείς ε, που θα συμμετέχουν εν πάση περιπτώσει στην υπηρεσία, τους εθνικούς εντεταλμένους εισαγγελείς, βλέποντας στο βιογραφικό σας ότι έχετε εργαστεί σχεδόν αποκλειστικά στη Ρουμανία ή επίσης σε κάποιες περιπτώσεις σε Μολδαβία και, και Μαυροβούνιο. Μπορείτε να μου απαντήσετε και ε, αγγλικά. Νομίζω ότι μπορούν να σας παρακολουθήσουν στη χώρα σας και μέσω των αγγλικών, λέει η κυρία Γιάλα Σέντερ. Θα υπερασπιστώ την ανεξαρτησία με βάση τα αποτέλεσμα που έχω πετύχει μέχρι τώρα. Μπορείτε να μιλήσετε ό,τι γλώσσα θέλετε, λέει η κυρία Κρέσλε. Δεν ξέρω αν θα ολοκληρώσω σε δύο λεπτά, αλλά θα απαντήσω. Πάντα ήμουν ανεξάρτητη. Σεβάστηκα πάντα την ομοθεσία. Τα αποτελέσματα που έχω πετύχει μιλούν από μόνα τους, διότι μαζί με τους συνεργάτες μου έχουμε ερευνήσει μέλη διαφόρων κομμάτων. Όχι όλα τα μέλη μια, ενός πολιτικού κόμματος. Επίσης, διενεργήσαμε έρευνες εις βάρος ανθρώπων πλούσιων σε σημαντικές θέσεις, αλλά επειδή ήμασταν ανεξάρτητοι, Πάντα ολοκληρώναμε τις υποθέσεις. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα να λέμε ότι η ανεξαρτησία παρέχεται, προβλέπεται από τον νόμο. Αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες για να περιοριστεί η ανεξαρτησία μας. Κατά τη γνώμη μας, ε, μια από τις προϋποθέσεις ε, για την ε, διενέργεια ερευνών για διαφθορά ή απάτη με οικονομικούς πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η προϋπόθεση είναι να είμαστε ανεξάρτητοι. Όσον αφορά το πώς ε, θα συνεργαστώ με άλλους Ευρωπαίους εισαγγελεί. Ήδη είπα ότι έχω συνεργαστεί με συναδέρφους από 40 διαφορετικά κράτη. Ήμουν εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Μαυροβούνιο, στη Μολδαβία διότι χρειάζονται τις εμπειρίες μας, τις πρακτικές μας και ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων μας, εγώ και οι συνεργάτες μου προσκληθήκαμε να, ως εμπειρογνώμονες για να εξετάσουμε την νομοθεσία. Συνεργαστήκαμε λοιπόν και με συναδέλφους μας στο πλαίσιο επαγγελματικών καταρτήσεων. Άνθρωπος είμαι, ε, αλλά αν δεν είμαι, αλλά ε, έχω τράξει σήμερα, διότι είναι πολύ σημαντική ημέρα σήμερα ε, και ε, και για, τους, ε, και για μένα και για τους συνεργάτες μου. Και μιλάω αγγλικά, αλλά γι' αυτό ήταν σημαντικό για μένα να μιλήσω ρουμάνικα. Αν θέλετε να σας μιλήσω μόνο αγγλικά, αλλά σας παρακαλώ καταλάβετε ότι και για μένα και για τους συναδέλφους μου είναι πολύ σημαντική η σημερινή μέρα. Η κυρία Μακοβέη, παρακαλώ. The people are talking. Monica, Monica has the floor. Η Μόνικα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συνεχίσω με βάση την ερώτηση που έθεσα ως μέλος της Επιτροπής ΕΛΥΜΠΕ. Τώρα μιλώ ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Είπαμε ότι γνωρίζετε τα βασικά χαρακτηριστικά των υποθέσεων απάτης. Μήπως όμως μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο παραπάνω γι' αυτό. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας τέτοια υπόθεσης και μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα των τρόπων με τον οποίο μπορεί ο Όλαφ να συνεχίσει τις εργασίες του πάνω στις παρατυπίες. Δεν είναι όλες οι παρατυπίες υποθέσεις απάτης. Και αναφέρομαι και στο ερώτημα της κυρίας Γκρέσλε. Ο Όλαφ θα μπορέσει να συνεχίσει να εργάζεται πάνω, να εξετάζει περιπτώσεις παρατυπίες. Όσον αφορά τις πιο συνηθισμένες υποθέσεις, μιλάμε για χρήση οικονομικών πόρων της Ένωσης για στόχους άλλους από αυτούς για τους οποίους προβλέπονται. Επίσης, διαφθορά όσον αφορά ευρωπαϊκούς πόρους. Είχαμε πολλές τέτοιες υποθέσεις στη Ρουμανία. Επίσης, έχουμε περιπτώσεις επιχειρήσεων ειδικευμένων στην ε, παραγωγή εγγράφων για ε, να υποβάλει κανείς αίτηση για να λάβει ευρωπαϊκούς πόρους. Είχαμε λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις, ε, είχαμε περιπτώσεις αξιωματούχων ε, που δέχονταν δωροδοκία ή άλλα πλεονεκτήματα για να ξεκινήσουν για να επιταχύνουν τις αιτήσει ή να ευνοήσουν αιτήσει ε, για ευρωπαϊκούς πόρους. Επίσης, είχαμε περιπτώσεις δικαιούχων ε, ευρωπαϊκών πόρων που χρηματοδότησαν ενδιάμεσες επιχειρήσεις που έτσι εμπόδιζαν άλλε επιχειρήσεις από το να λάβουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Όσον αφορά τον Όλαφ, πράγματι δεν είναι όλε οι υποθέσει περιπτώσει απάτης. Υπάρχουν αρκετές που αφορούν απλά παρατυπίε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να μπορεί να διαβιβάζει μια υπόθεση στον Όλαφ και να βρίσκεται σε επαφή και με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Η κυρία Κρίσμπεκ, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα ε, να βγω λίγο από την σημαντική βεβαίω συζήτηση ε, σχετικά με την ε, δυσκολία που έχετε αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια για να διαφυλάξετε την ανεξαρτησία της αρμοδιότητός σας για να επανέλθω στα του γραφείου της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Εμείς, η δική μας πολιτική ομάδα, πάντοτε είμαστε υπέρ της αποκεντρωμένης ε, δομής και της Ευρωπαϊκής εισαγγελία που θα έχει μια μεικτή δομή ως προς το θέμα της αποκέντρωσης. Πώς βλέπετε εσείς ε, την ε, λειτουργία της και ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών αλλά και της ομαλής του λειτουργίας ως προς ακριβώς τα θέματα κεντρι, κεντρικοπαγούς και αποκεντρωμένης δομής που και τα δύο θα πρέπει να ενέχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κοιτάξτε, θα είναι μια πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ή ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής εισαγγελία. Η εισαγγελία συνήθως ε, λειτουργεί ως ενιαία ε, ε, ομάδα και εγώ έτσι έδρασα, αλλά η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει κάποια πλέον εκτήματα, έχει κάποια μόνιμα σώματα και εγω ετσι εδρασα αλλα η υπηρεσια της ευρωπαικης εισαγγελιας εχει καποια πλεονεκτήματα, εχει καποια μονιμα σωματα και εχει και κάποιους ε, εν πάση περιπτώσει απεσπασμένους εισαγγελεί, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία με τις εθνικές εισαγγελίε. Ε, θα είναι σημαντικό να έχουμε ομαλή συνεργασία με αυτές αλλά και θα είναι ακόμα πιο σημαντικό να έχουμε έναν εσωτερικό κανονισμό, κανόνες, διατάξεις που θα διέπουν με απόλυτη ε, με συγκεκριμένο τρόπο την δουλειά μας και την εντολή μας και θα πρέπει να έχουμε και ένα case management system, δηλαδή ένα σύστημα διαχείρισης φακέλων που θα μας επιτρέπει να, να εντοπίζουμε κάθε φορά ποιες είναι οι επαφές που είχαμε με ποιους δικαστικούς λειτουργούς και για ποιο φάκελο. Οι ανταλλαγές μεταξύ των ε, γραφείων της αγγελίας μπορούν να γίνουν πολύ γρήγορα ε, σε θεσμικό ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της EPPO, της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, για την έναρξη ερευνών, για παράδειγμα, εντός τριών ημερών που είναι μια τέτοια προθεσμία για την τέτοια απόφαση, είναι ο χρόνος ε, ε, ανταπόκρισης της ε, είναι πολύ γρήγορος. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε λέει ο κύριος Ζάβορ, ευχαριστώ την κυρία Κιόβεση που είναι πάλι μαζί μας εδώ. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα ε, που έθεσε η κυρία ε, ε για τις απάτες ε, των ευρωπαϊκών πόρων που πολύ συχνά λαμβάνουν χώρα σε πολλές ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Εσείς προερχόμενοι από την περιοχή αυτή και έχοντας μια τεράστια εμπειρία για την αντιμετώπιση της συστημικής ε, διαφθοράς και γνωρίζοντας ε, τι πρέπει να γίνει όταν πολιτικές πιέσεις, ακόμα και κυβερνήσεις ή και κάποιες ε, ομάδες της μαφίας κινούνται για να ασκήσουν την επιρροή τους. Εσείς Πώς νομίζετε ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε τη δική σας εμπειρία ώστε η Ευρωπαϊκή ε, Εισαγγελία να είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τα υφιστάμενα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, δεν πρέπει κανείς να έχει προκατασκευασμένες ιδέες. Ε, εγώ αν ήμουν επικεφαλής της Τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έβλεπα ότι μία χώρα θα είχε περισσότερες απάτες από άλλη, αν αυτό μου το έδειχναν οι στατιστικέ. τι να σα πω, για περιπτώσεις που δεν έχουν ερευνηθεί και που δεν έχουν αποδεχθεί δεν λέει και πολλά. Ε, σε, σε άνω των 2.000 ε, ετήσιων περιπτώσεων, το να έχω μάλλον εξετάσει άνω των 2.000 περιπτώσεων ε, ε, απάτηση με ευρωπαϊκού πόρου, μου δίνει μια μεγάλη εμπειρία αλλά ο τρόπο με τον οποίο γίνονται οι απάτες αυτέ, ε, μεθοδολογικά είναι αρκετά παρόμοιο. και επομένω αυτό πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αναπτύξει μεθοδολογίε αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. Εσείς αναφερθήκατε στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Αν δείτε την έκθεση της Όλαφ θα δείτε τι συμβαίνει ε, σε σχέση με ε, στοιχεία που έχουν αποδειχθεί από την Όλαφ. Βλέπουμε όμως ότι, ε, ε, ότι υπάρχει μια τάση να γίνεται συστημική πλέον η διαφθορά, η απάτη των ευρωπαϊκών πόρων και επομένως η αρμοδιότητα της εισαγγελίας δεν είναι μόνο να ερευνά περίπλοκες ε, περιπτώσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ αλλά να ερευνά και εκείνες περιοχές, εκείνα τα πεδία που λαμβάνουν χώρα οι απάτες κατ' ακόμα και αν αφορούν μικρά σχετικώς ποσά. Νομίζω ότι αυτό που η d στη Ρουμανία έκανε ήταν αυτό τα τελευταία χρόνια και αν δείτε τα αποτελέσματα που επιτύχαμε ήταν απολύτως σχετικά με τις απάτες των ευρωπαϊκών πόρων. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη εμπειρία. Θα μπορούσε να κινητοποιηθεί για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Direkt dahinter, Kollege bitte. Ο συνάδελφος ο Μάτζη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρία Κιόβεση, έχετε ήδη απαντήσει πάρα πολλά ερωτήματα. Ήθελα να σας πω ότι είμαστε πολλοί εδώ που δεν δίνουμε καμία σημασία σε αυτήν την εκστρατεία που θέλει να ε, επιχειρεί να σπηλώσει το όνομά σας. Είμαστε απολύτως πεπισμένοι για το θάρρος σας. Και πιστέψτε με, σε πολλές άλλες χώρες είχαμε τέτοιες επιθέσεις κατά προσώπων, ιδιαίτερα ε, εισαγγελέων και δικαστικών λειτουργών. Και υπάρχει μια ομοιότητα σε όλες τις χώρες. Όταν ο δικαστικός λειτουργός ή ο εισαγγελέα κάνει καλά τη δουλειά του, ξαφνικά του απευθύνονται κατηγορίες και του ασκούνται πιέσει. Λοιπόν, τώρα σχετικά με τους ε, ε, whistleblowers ε, σχετικά με αυτούς που καταγγέλνουν περιπτώσεις απάτης και εγκληματική δραστηριότητα. Ήθελα να μου πείτε ε, κατά πόσον θεωρείτε ότι αυτοί οι whistleblowers θα πρέπει να προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι αυτό το τμήμα του κειμένου, σας κάνω την ερώτηση, διότι το σχετικό τμήμα του κειμένου δεν έχει ακόμα φτάσει προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Ehm, γνωρίζω την ε, έννοια πράγματι των πληροφοριοδοτών. Η Ρουμανία έχει περάσει ειδική νομοθεσία ακριβώς για το θέμα και υπάρχουν και κάποια μέτρα προστασίας τους και σαφείς ε, κανόνες. Ε, κοιτάξτε, λειτουργεί το σύστημα αυτό στη Ρουμανία. Η απόφαση όμως να περάσει μια τέτοια οδηγία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Εγώ μπορώ να σας δώσω την απόψή μου ως εισαγγελέα, αλλά είναι κάτι το οποίο λαμβάνει ως απόφαση ο συνομοθέτης. Έχουμε μια η ειδική ε, νομοθεσία και στην ΔΕΝΑ ε, επίσης εργαζόμαστε με τέτοιους ε, πληροφοριοδότες. Κυρία Πιτέρα. <clears throat> Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα που αφορά το πλαίσιο αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ε, Θεωρείτε ότι τα προνόμια και οι αρμοδιότητες ε, επαρκούν για να διώξει επαρκώς ε, το οικονομικό έγκλημα. Necesitatea de a Η ανάγκη έγκρισης αυτού του κανονισμού και δημιουργίας ενός γραφείου Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρεται στο άρθρο 83 της συνθήκης, αν δεν κάνω λάθος, αλλά θα επανέλθω. Η απόφαση η επέκταση των αρμοδιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Αγγελία είναι μια απόφαση που θα λάβουν οι συνομοθέτε. Είναι δύσκολο να πούμε τώρα ότι ναι, αυτό πρέπει να γίνει και να διευρυνθούν οι αρμοδιότητε. Εάν δείτε, παραδείγματο χάρη, την απάτη που περιλαμβάνει ευρωπαϊκά κονδύλια χρηματοδότηση, παραδείγματο χάρη ε, τρομοκρατικών πράξεων, τότε θα έλεγα ότι ναι, σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται. Αν δούμε όμως την προστασία άλλων αξιών θεμελιωδών, τότε θα έλεγα ότι α, αυτή τη στιγμή ας δούμε αν λειτουργεί και μετά θα λάβουμε μια απόφαση. Αλλά ούτω ή άλλω είναι μια απόφαση που επαφίεται στου συνομοθέτες. Αυτό το οποίο θα έκανα εγώ θα ήταν να αναλύσω τα μοτίβα του εγκλήματος, το πώς εμφανίζονται και να δω την πιθανή σχέση με οικονομικά εγκλήματα και άλλα σοβαρά εγκλήματα όπως το οργανωμένο έγκλημα και την ε, τρομοκρατία. Και αν δείτε ότι εκεί πέρα υπάρχει μία ανάγκη διεύνησης των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής αγγελίας. Ε, τότε εκείνη τη στιγμή θα μπορέσουμε να αποστείλουμε την ε, γνωμοδότησή μας ε, στους συνομοθέτες. Δεν νομοθετούμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προσφέρουμε την ε, τεκμηριωμένη γνώμη μας, ειδικά αν πρόκειται για νομοθεσία η οποία εμποδίζει την δουλειά μας ως εισαγγελής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση, τον χρόνο που μας αφιερώσατε. Ευχόμαστε καλή τύχη. Ε, θα συνεχίσουμε εμείς μετά το τέλος συνεδρίασης. Συναδελφοί, λίγο την υπομονή σας θα εξηγήσω λίγο την διαδικασία. Να ευχαριστήσω την κυρία Κοβέση πρώτα απ' όλα για τη συμμετοχή της. Ε, συναδελφοί, ένα λεπτό. θα γίνει μια πλήρης αξιολόγηση της ακρόασης ε, και όπως με όλους τους υποψηφίους θα αποστείλω μια επιστολή στον πρόεδρο Ταγιάννη που θα παρουσιάσει την θέση μας και την θέση της Επιτροπής Ελέγχου ε, του Προπολογισμού όπως θα μου τη διαβάσει η κυρία Γκρέσλε. Σας ευχαριστώ εξ ονόματος Επιτροπής μας ε, και θα κάνω τώρα κάποιες ανακοινώσεις, εσείς μπορείτε να φύγετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι,